Right, Ας ξεκινήσουμε για να μην χάνουμε χρόνο και θα ήθελα να σας πω, αναλαμβάνοντας την Προεδρία, ότι χαίρομαι που μπορώ να προεδρεύσω αυτόν τον δύο συνεδριάσεων. Το έχω πράξει και στο παρελθόν, αλλά πρόκειτο μόνο για το Κορεπέρ και υπήρχαν μόνο 12 κράτη, άρα δεν ήταν τόσο σημαντικό. Αλλά ε, το να υπάρχει ένας βουλευτής στην, ε, ε, σαν πρόεδρος αυτής της συνεδρία είναι πολύ σημαντικό και σημαδιακό, διότι δείχνει ότι υπάρχει μία μία ευθύνη η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται και να αναλαμβάνεται και από τα εθνικά κοινοβούλια και θα πρέπει να συνεργαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα εθνικά κοινοβούλια για να υπάρχει μία συστηματική εποπτεία και παρακολούθηση των οργανώσεων τα οποία πρέπει να παρακολουθούν από κοινού τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε σήμερα το πρωί δύο συνεδριάσεις. Το πρώτο μέρος, το οποίο θα ξεκινήσει τώρα, αναφέρεται στην προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και της συνεργασίας του Σέιγγεν και θα εξετάσουμε τον ρόλο του, της Frontex, διότι ο πρόεδρος της κάθεται αριστερά μου. Και μετά στις 10.30 θα έχουμε τη συνεδρίαση λήξη η οποία περιγράφεται ε, ως ε, ε, συνοπτική δηλαδή πώς θα γίνει ένα αρμονικό συντέριασμα με ποιους τρόπους μπορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ισχύσουν την κοινή του συνεργασία και εποπτεία των οργανισμών. Έχουμε τρεις ομιλητές τώρα στο πρώτο μέρος, τον κύριο Λέιτινεν, ο κύριος Μπουσουτήλ, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει μπλοκάρει στην κίνηση και ελπίζω ότι θα έρθει γρήγορα η κίνηση γητή σχετικά με το, την Frontex ή ε, τον ε, στην Επιτροπή Ελευθεριών και την κυρία Τσόνογλου που είναι εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και θα δώσω τον λόγο ε, στη συνέχεια ε, για ερωτήσεις σε δύο εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και έναν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ούτω καθεξής και ελπίζω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τις 10.30 αυτό το τμήμα και αυτές οι παρεμβάσεις παρακαλώ να μην ξεπεράσουν δύο λεπτά από το κοινό για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο στους περισσότερους δυνατούς. Τώρα λοιπόν δίνω το λόγο καταρχήν ή στο Διευθυντή του Frontex ο οποίος θα παρουσιάσει και μία προβολή PowerPoint και έτσι θα παρακολουθείτε αυτά τα οποία λέγει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας. Και πάλι είναι τιμή μου να παρευρίσκομαι στην κοινή συνεδρίαση, στη μεικτή συνεδρίαση Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Στα επόμενα δεκαλεπτά λεπτά θα σας ε, εξηγήσω ή θα σας επενθυμίσω το πεδίο, το σκοπό της, ε, του ελέγχου των συνόρων από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά και θα τονίσω ορισμένα θέματα που σχετιζόνται με τη Frontex και το συνοριακό έλεγχο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο σύνολό του. Το πρώτο που θέλω να δούμε είναι οι κύριοι στόχοι. Νομίζω ότι είναι δυτή. Εμείς ασχολούμαστε με τη διαχείριση των συνόρων αφενός και αφετέρου με την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου κλίματος στα σύνορα. Ο κύριος στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι στα σύνορα γίνονται σεβαστοί οι κανόνες, αλλά ο στόχος μας είναι επίσης να διασφαλίσουμε τις ε, νόμιμες και ομαλές συνοριακές, διασυνοριακές δραστηριότητες. Φυσικά, η προσέγγιση μας είναι ευρωπαϊκή, καθώς έχουμε την ευρωπαϊκή πολιτική, έχουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το συνοριακό έλεγχο, και πρέπει να διαφυλάξουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα από τα κύρια από τα θεμελιώδη δικαιώματα σήμερα και πρέπει να γίνεται σεβαστή. Αυτή είναι η στόχη λοιπόν. Επόμενη διαφάνεια. Θέλω να σας υπενθυμίσω επίσης ε, την ε, στρατηγική, την ολοκληρωμένη στρατηγική συνολικής ασφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε πέντε κυρία στοιχεία. Τα πρώτα στοιχεία να κάνουν ε, με όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του νόμου και το με όσους αποφασίζουν, νομοθετούν. Επίσης ε, έχουμε τους συνοριακούς ελέγχους, την εποπτεία των συνόρων, έχουμε όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ε, για να ανοιχνεύσουμε και να εντοπίσουμε το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα στα σύνορα. Το τρίτο στοιχείο είναι η γεωγραφική εμβέλεια των δραστηριοτήτων μας, δηλαδή θέλουμε να δρούμε όχι μόνο στα σύνορα αλλά πριν, ε, επί των σύνορων και πίσω από τα σύνορα. Και το τέταρτο στοιχείο έχει να κάνει με την δύο οργανική συνεργασία μεταξύ των οργανισμών. Εδώ μπορούν να υπάρξουν πολλές βελτιώσεις, δηλαδή να συνεργάζονται οι αρχές που δραστηριοποιούνται στη σύνορα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και επίπεδο και διεθνές επίπεδο. Κάτι, όπως σας είπα, το τελευταίο στοιχείο έχει να κάνει με τους νομοθέτες. Δηλαδή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πολιτικό πλαίσιο είναι παρκές ε, προκειμένου να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας. Τώρα, να περάσουμε στο ρόλο της Frontex. Δεν θα σας απαριθμίσω τα νομικά καθήκοντα, αλλά θα προσπαθήσω να σας περιγράψω ποιος είναι ο ρόλος μας. Το Σημείο φετηρία είναι ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αναφέρεται ρητά στη συνθήκη τη Λισαβόνα, Αυτή η προσέγγιση υπάρχει παντού και στο πρόγραμμα τη Στοκόλμη, τη στρατηγική εσωτερική ασφάλειας, παντού. Και αυτό ο επιμερισμό ευθυνών είναι κάτι μη αμφισβητήσιμο. Αυτό σημαίνει ότι η Frontex δεν είναι ο οργανισμό ο οποίος λαμβάνει τι αποφάσει εκ μέρου των κρατών μελών. Πάντοτε τα κράτη-μέλη είναι αυτά που λαμβάνουν τις αποφάσεις, χορηγώντας την είσοδο και τα συνεπακόλουθα. Ο δικός μας ρόλος είναι να προσθέσουμε αξία στις επιδόσεις των κρατών μελών, στις πράξεις των κρατών μελών και γι' αυτό έχουμε ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο στη διάθεσή μας. Είμαστε ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, προωθούμε την ευρωπαϊκή πτυχή, γι' αυτό ιδρυθήκαμε προωθούμε τον ε, ευρωπαϊκό πολιτισμό φύλαξη των συνόρων. Αυτό συνίσταται στο πώς θέλουν οι Ευρωπαίοι να ελέγχουν τα εξωτερικά σύνορα. Ξεκινώντας από μία από τις ε, κύριες αξίες που είναι ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, προσπαθούμε να έχουμε περαιτέρω εναρμόνιση και διαλειτουργικότητα γιατί μόνο αν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιους ε, εναρμονισμένους τρόπους δράσης, μόντιο ε, περάντη, και με την κατάλληλη κατάρτιση, τότε μόνο τα κρατημέλη μπορούν να ελέγξουν τα σύνορα. Έτσι λοιπόν ο στόχος είναι να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε τις επιδόσεις των κρατών μελών. Αυτός είναι ο ρόλος της Frontex. Έχουμε ένα μέσο για να, να ευαισθητοποιούμε τα κράτη-μέλη για την κατάσταση. Έχουμε ένα πλήρες δίκτυο αναλυτικών ικανοτήτων και τα κράτη-μέλη γνωρίζουν πώς έχει η κατάσταση και επίσης κάνουμε και προβλέψεις για το μέλλον. Αυτή είναι η προσθετή αξία μας. Ένα άλλο ε, τμήμα των καθηκόντων μας ε, είναι η εκπόνηση πιλωτικών ε, προγραμμάτων και οι κοινέ επιχειρήσεις. Είχαμε κοινή επιχείρηση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη Μεσόγειο, στα Κανάρια, στα αεροδρόμια και επιχειρήσεις επιστροφών. Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα τμήματα των δραστηριοτήτων μας, αλλά ο στόχος αυτών των κοινών επιχειρήσεων δεν είναι να αντικαταστήσουμε τις ε, εθνικές ικανότητες, αλλά να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε την ικανότητα του κράτους μέλους. Σε κάθε επιχείρηση το κάθε... ο στόχος είναι να ενισχύσουμε την ικανότητα της χώρας να ελέγξει τα σύνορά της. Ένα πρόσθετο στοιχείο ε, είναι η κατάρτιση και η έρευνα. Εδώ έχουμε ήδη συστήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη για το συνεργειακό έλεγχο σήμερα. Εργαζόμαστε σε ε, προγράμματα ενδιάμεσοπιπέδου και επίσης ε, τώρα εκπονούμε και προγράμματα για τριτοβάθμια εκπαίδευση για να ενδυναμώσουμε τους συνορικούς ελέγχους. Κατόπιν, ικανότητα της Frontex, εμπειρογνωμοσύνη. Έχουμε προσωπικό 300 ατόμων. Αυτούς τους ανθρώπινους πόρους. Έχουμε αυτόν το προσωπικό μας. Έχουμε αναλυτικές ικανότητες, έχουμε τη μεθοδολογία να εφαρμόσουμε συστηματικά τις πληροφορίες που έχουμε λάβει κυρίως από τα κράτη-μέλη αλλά και από άλλες πηγές ε, όπως από το ε, κοινό μοντέλο, ολοκληρωμένο μοντέλο ανάλυσης κινδύνου και ε, το τι προκύπτει από τις αναλύσεις αυτές δίνονται στα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η γνώση τους για να ευαισθητοποιηθούν. Επίσης, ε, έχουμε τις ευρωπαϊκές ομάδες σύνοριοφυλάκων και έχουμε και μία σειρά τεχνικών μέσων, σκάφη, ελικόπτερα κτλ. Και με το νέο τροποποιημένο μενοκονισμού θα έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε δικό μας εξοπλισμό. Και πάλι πώς θα το πράξουμε και γιατί το πράττουμε. Αυτό η πράξη μας ακολουθεί τις ανάγκες. Και έχουμε και τον προϋπολογισμό που έχει ως στόχο να αντισταθμίσει την συμμετοχή των κρατών μελών στις κοινέ επιχειρήσεις που οργανώνουμε, που συντονίζουμε εμείς. Στη συνέχεια να σας πω δύο λόγια για το μέλλον. Ανέφερα ήδη τον τροποποιημένο κανονισμό που θα τέθει σε ισχύ πολύ σύντομα και αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική της Frontex θα πρέπει αναλόγως να τροποποιηθεί. Ο κανονισμός φυσικά είναι το σημείο φετήριας, αλλά ένας άλλος στρατηγικός παράγοντας είναι το πρόγραμμα που τρέχει σήμερα από την Κομισιόν. Πρόκειται για το σύστημα Eurosur, το σύστημα εποπτείας. Αυτό θα γίνει ένα κύριο μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με τη Frontex ε, στον τομέα των συνοριακών ελέγχων. Και φυσικά πρέπει να δεκτούμε και τα γεγονότα. Πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με το τι συμβαίνει στον οικονομικό τομέα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα σύστημα καλύτερων δικτών ε, για τις επιδόσεις μας και πρέπει να δούμε που μπορούμε ε, να βελτιώσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Σίμων Μπουζουτήλ όπως σας είπα και πριν είναι εισηγητής για το νέο κανονισμό του Frontex. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζω ζητώντα συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Είχα πέσει σε μποτιλιάρισμα. Ως Ευρωβουλευτής πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα που θέτει το θέμα μας, δηλαδή τι είναι η δημοκρατική λογοδοσία για, αυτό, για αυτή την υπηρεσία. Πολύ. πολύ υπέβαλαν δύο κατηγορίες παραπώνων και προσφυγών από τη μία άνθρωποι που προέρχονται από χώρες που υφίστανται μεγάλες μεταναστευτικές ροές θεωρούν ότι δεν είναι αποτελεσματική η υπηρεσία. Από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι αυτή η υπηρεσία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τουλάχιστον κλείνει τα μάτια στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και οι δύο αυτές κατηγορίες είναι σοβαρές και πρέπει να τις συζητήσουμε. Αυτό είχαν κατά νου και οι ευρωβουλευτές που πρόσφατα ενέκριναν την αναθεώρηση του κανονισμού με τη νέα εντολή της υπηρεσίας. Βασικά απαντήσαμε ότι βεβαίως πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, να γίνει πιο αποτελεσματικός, πιο ορατός αλλά επίσης να ενδυναμώσουμε την λογοδοσία του. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας αναφέρω μερικούς τρόπους με τους οποίους ελπίζουμε να αυξηθεί η δημοκρατική εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής από τώρα και στο εξής. Γιατί θεωρούμε ότι έτσι απαντάμε στις δύο ανησυχίες που εξέφρασα προηγουμένως, δηλαδή αποτελεσματικότητας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, η δημοκρατική εποπτεία, για τη δημοκρατική εποπτεία με τις τροπολογίες του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε, ανταποκρίθηκε, ζήτησε τις αλλαγές που θα σας απαριθμίσω τώρα ως βελτίωση της λογοδοσίας της υπηρεσίας αυτής. Βάλαμε στο νομοσχέδιο μία ρήτρα που αναφέρει ότι ο αριθμός των υπεύθυνων για τους ελέγχους στα σύνορα θα δημοσιεύεται τακτικά και ότι οι πληροφορίες αυτές τώρα νομικά θα υποχρεωτικά θα υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές εγκαταστάσεις που διαθέτει κάθε χώρα μέλος προς την υπηρεσία. Ξέρετε ότι για ορισμένα χρόνια η υπηρεσία αυτή αντιμετώπιζε δυσκολίες να, να εφαρμόσει την εντολή της. Γιατί έπρεπε τα κράτη-μέλη να χορηγήσουν τους ανθρώπινους πόρους και τις εγκαταστάσεις, τα ελικόπτερα, τα πλοία κλπ. Και οι χώρες μέλη δεν το έπραταν. Ε, είχαν υποσχεθεί ότι θα χορηγήσουν τέτοιους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, αλλά όταν έφτανε ο κόμπος στο χτένι δεν το έπραταν. Επομένως, ένας τρόπος να τους υποχρεώσουμε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αυτές είναι αυτή η ρήτρα που στο εξή υποχρεώνει την υπηρεσία να δημοσιεύει τακτικά τι χορηγεί το κάθε κράτος μέλος. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο αυξάνουμε την δημοκρατική εποπτεία είναι να διασφαλίζουμε ότι όλες οι συμφωνίες που συνάπτει με άλλες υπηρεσίες όπως για το άσυλο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή και για την Ευρωάστα θα γνωστοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί αυτό το τελευταίο να ασκεί μια μεγαλύτερη εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής και ως προς τη συνεργασία της με άλλες. Επίσης, θα πρέπει τώρα να χορηγεί πληροφόρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για συμφωνίες που συνάπτει με τρίτες χώρες. Αυτό είναι μεγάλο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί δεν ξέρουμε πάντοτε ποιες συμφωνίες συνάπτει η υπηρεσία με τρίτες χώρες, ποιες χώρες με ποιες χώρες είναι σε θέση να συνάψει συμφωνίες, ποιες χώρες έχουν ανεπαρκή σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επίσης θα είναι υποχρεωμένη να πληροφορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την για τον ορισμό συνδέσμων σε τρίτες χώρες. Είχα πει και από την αρχή ότι από, τα μεγάλη, από τις μεγαλύτερες κατηγορίες που αντιμετώπισε, παράπονα που αντιμετώπισε η υπηρεσία είναι ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, ας πούμε, αφήνουν ανθρώπους να πνιγούν στη θάλασσα. Αυτό είναι πολύ σοβαρή κατηγορία, πράγματι. Και εγώ δεν συμμερίζομαι την ανησυχία αυτή, γιατί νομίζω ότι τέτοιου είδους φαινόμενα ε, καλύπτονται από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι έπρεπε να τις αντιμετωπίσουμε και τις αντιμετωπίσαμε ως εξής. Δημιουργήσαμε ένα μηχανισμό επιτήρησης ή εποπτείας που να εξετάζει, να παρακολουθεί τις δραστηριότητες όλων των σχετικών υπηρεσιών από απόψεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα υπάρχει στο εξής ένας ειδικός αξιωματούχος για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην υπηρεσία που θα δρά ανεξαρτήτως από τους άλλους. Και θα καθοριστεί, θα οριστεί επίσης ένα συμβουλευτικό σώμα, ένα συμβουλευτικό βήμα που να ενημερώνει και με άλλες υπηρεσίες όπως την υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για να παρατηρεί κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν η υπηρεσία ή παρατηρήσει οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια της αποστολή, τότε για πρώτη φορά προβλέπεται ακόμη και η δυνατότητα να αρθεί, να τερματιστεί κάποια αποστολή. Αυτό νομίζω ότι απαντάει όντως επαρκώς στις ανησυχίες για θεμητές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά βέβαια απαιτεί έναν σοβαρό μηχανισμό εποπτείας. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους θεωρούμε ότι έχει διασφαλιστεί η εποπτεία όπως στην περίπτωση διεκπαιρέωσης των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατόμου κατά τη διάρκεια μιας αποστολής πρέπει η υπηρεσία να σέβεται αυστηρά ό,τι ισχύει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η καινούργια ρήτρα διατυπώθηκε σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων. Και έτσι διασφαλίσαμε επίσης ότι και από αυτή την άποψη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων οι δραστηριότητες της υπηρεσίας δεν θα δημιουργήσουν στο, δημιουργούν στο εξής τέτοιες ανησυχίες. Τώρα για τις ε, επιστροφές μεταναστών στη χώρα προέλευσης. Και αυτό ήταν με ανησυχία πολλών. Εάν επιστρέφονται άνθρωποι στην χώρα προέλευσής τους, υπάρχει καμία επιτήρηση ως προς το πώς γίνεται αυτό. Από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποια είναι η τύχη τους αφού επιστραφούν. στο νομοσχέδιο βάλαμε μια ρήτρα που λέει ότι σε αιτήσια βάση η Επιτροπή Κομισιόν πρέπει να αναφέρει η Κομισιόν, όχι πια η ίδια υπηρεσία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι εποπτεία έχει γίνει για την τύχη των ανθρώπων αυτών από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Δηλαδή στο εξής, όλες οι επιχειρήσεις επιστροφής μεταναστών θα παρακολουθούνται. Αυστηρά από την Κομισιόν η οποία με τη σειρά θα πρέπει να μας πληροφορεί εμάς πώς και αν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και βέβαια μπορούμε να προσκαλούμε τον Διευθυντή της Υπηρεσίας τακτικά στο Κοινοβούλιο. Όσες φορές του το ζητήσαμε το έπραξε προθήμως και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τέλος, για τον προϋπολογισμό, είναι γνωστό ότι αν δεν έχει κανείς πόρους δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε μέγας σύμμαχος της υπηρεσίας διασφαλίζοντας ότι θα έχει ό,τι πόρους χρειάζεται γιατί ως τμήμα της αρχής ε, για τον προϋπολογισμό το Κοινοβούλιο αύξησε τον λειτουργικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας για να της επιτρέψει να πράξει ό,τι πρέπει να πράττει. Ελπίζω να έχετε έτσι μια γενική ιδέα των επιχειρημάτων μας και των τρόπων με τους οποίους θελήσαμε να λύσουμε τα προβλήματα που είχαν αναφερθεί. Τώρα βέβαια πρέπει να αντιδράσει η ίδια η υπηρεσία ώστε ο κανονισμός αυτός μόλις θεθεί ενισχύ να εφαρμοστεί κιόλα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή Ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ χρήσιμη επισκόπηση και η τρίτη ομιλήτρια είναι η κυρία Βασιλική Τσονογλού η οποία θα μιλήσει σαν μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία υπέφερε πάρα πολύ από την ε, μεγάλη αύξηση της ε, λαθρομετανάστευσης Έχετε το λόγο. Αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για μένα, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να σας μιλάω για ένα τόσο σημαντικό για τη χώρα μου ζήτημα η ελλάδα όπως και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου πλήττεται σοβαρά από τις δυσανάλογες μεταναστευτικές ροές στα εξωτερικά της σύνορα. τα εκτεταμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και η εγκύτητά της με τις χώρες διέλευσης και καταγωγής παράνομων μεταναστών την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη. και επειδή οι αριθμοί είναι κάποια φορά πολύτιμοι σύμμαχοι των λέξεων σας αναφέρω ενδεικτικά ότι μόνο πέρυσι το προηγούμενο προηγούμενο έτος συνελήφθησαν στη χώρα μας χιλιάδες παράνομοι μετανάστες κατά το τρέχον έτος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην ελλάδα 43.859 μη νόμιμοι μετανάστες αριθμός μειωμένος κατά 39,31% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010 ωστόσο σε καμιά περίπτωση καθησυχαστικός. οι πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στην βόρεια αφρική επιβαρύνουν σημαντικά τους παράγοντες δημιουργίας μεταναστευτικών ροών προς την νότια ευρώπη και τους καλούν σε εγρήγορση το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα. αποτελεί καταρχήν ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. οι ελληνικές αρχές διαχειρίζονται στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα χιλιάδες ψυχές μεγέθη που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους. καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αγωνία και την ελπίδα των μεταναστών για μια καλύτερη ζωή αλλά και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας σε συνθήκες δύσκολες. Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί ζήτημα ασφάλειας για τη χώρα μας, που αφορά την υπονόμευση της κοινωνικής ειρήνης, της κοινωνικής σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής είναι εξαιρετικά δυσχερείς και κοστοβόρες οι συνθήκες στη διεκπαιρέωση αιτήσεων ασύλου και επαναπατρισμού βεβαίως στις χώρες τους των παρανόμων αυτών μεταναστών. Η παροχή ασύλου είναι ένα ζήτημα για το οποίο ασκείται συχνά εντονότατη κριτική στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου όμως να σας θέσω τον εξής προβληματισμό. Καταρχήν η κριτική είναι δίκαιο να ασκείται υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ισότητα σε ό,τι αφορά τους όρους μετανάστευσης στα κράτη-μέλη, γεγονός που επηρεάζει μοιραία και τους όρους του ασύλου όταν καλείται κανείς να εξετάσει χιλιάδες καταχρηστικές στη συντριπτική τους πλειοψηφία αιτήσεις ασύλου, τότε μοιραία ο χρόνος χάνεται και είναι σημαντικός. Το Εθνικό Σύστημα Ασύλου δέχεται σημαντικές πιέσεις. Για να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία του, εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης για την μεταρρύθμισή του, σε νομοθετικό κυρίως επίπεδο. Ωστόσο, οι προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικασιών ασύλου και των συνθηκών συνθηκών διαβίωση των ετούντων άσυλο στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσουν εάν παράλληλα και συμπληρωματικά δεν συγκροτηθεί ένας κοινό ευρωπαϊκός βηματισμός, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Το βάρος θα πρέπει να ανακατανεμηθεί με βάση πληθυσμιακά, οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια. Η αναθεώρηση του κανονισμού όπως Δουβλίνο 2 και ιδιαίτερα της αρχής της αποκλειστικής αρμοδιότητας του κράτους πρώτης παράνομης εισόδου είναι και δίκαιη και επιβεβλημένη. Στην παρούσα του μορφή ο κανονισμός επιβαρύνει υπέρμετρα και δυσανάλογα τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα τα οποία ως εκ της γεωγραφικής τους θέσεως καλούνται να εκτελέσουν τα καθήκοντα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν σύνολο. Είναι οξύμορο, είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε κριτική να προσάπτεται αυτός ο ψόγος για την Ελλάδα αυτή η κατηγορία. Και χωρίς να διεκδικούμε στη χώρα αυτή την πατρότητα όλων των θεσμών, ενδιαφέρον θα είχε κανείς να μελετήσει τις ρίζες του θεσμού που ανατρέχουν στην αρχαία Ελλάδα. Ο Έλληνας τραγωδό Εσχύλος καταγράφει στην πρώτη σωζόμενη τραγωδία του ακριβώς παράνομο ε, ε, ζήτημα, υπερβολικό ζήτημα μεταναστών τη εποχή εκείνη στο έργο του «Οικέτιδες». Ίσως με έκπληξη έκπληξη να διαπιστώνεται ότι το θέμα αυτό τόσο επίκαιρο αλλά και τόσο παλιό έχει τις ρίζες του στην ελληνική πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα να σας δώσω μια εικόνα της κατάστασης στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι όμως και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή από μόνη της η διαπίστωση αρκεί για να αποδείξει ότι το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί μόνο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό πρόβλημα και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η συνδρομή του frontex στην προσπάθεια των ελληνικών αρχών είναι κρίσιμη το κεκτημένο του σέγγεν προβλέπει την ενδυνάμωση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ευρωπαϊκής ένωσης. συνεπώς εκεί θα πρέπει να δοθεί και το βάρος για την αντιμετώπιση των τυχών ελλείψεων δηλαδή στην καλύτερη αστυνόμευσή τους με σκοπό την αποτροπή των παράνομων εισόδων. ο στόχος αυτός μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί μέσω της ενίσχυσης του ρόλου του frontex η κοινή επιχείρηση ποσειδών που διεξάγεται από το 2006 στα χερσαία και θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύνορα έχει αποδώσει καρπούς πράγματι. το επιχειρησιακό γραφείο του frontex στον πειραιά που λειτουργεί πιλωτικά με στόχο την ενίσχυση και την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής ικανότητας του οργανισμού στην περιοχή της νοτιοανατολικής μεσογείου αξιολογείται θετικά η ελλάδα επιδιώκει την μονιμοποίηση της λειτουργίας του μηχανισμού αυτού του προγράμματος αυτού. επίσης στηρίζουμε την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τόσο στον τομέα της αποτροπής εισόδου παράνομων μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και της άμεσης επιστροφής στην πατρίδα τους θα πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση στο ζήτημα των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στα κράτη μέλη αλλά η απομάκρυνσή τους δεν είναι εφικτή για τεχνικούς ή άλλους λόγους. η σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής είναι ένα πρακτικό πράγματι εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. τόσο όμως η κοινοτική πολιτική εθελούσιων και αναγκαστικών επιστροφών όπως και η άμεση προώθηση και ουσιαστική εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής θα πρέπει να ενταχθούν και αυτές στο συνολικό πλέγμα των σχέσεων της ένωσης με κάθε τρίτη χώρα. η ευρωπαϊκή ένωση είναι σε θέση να ασκήσει τις κατάλληλες πιέσεις και να παράσχει τα απαιτούμενα κίνητρα προς τρίτες χώρες προκειμένου να συνεργαστούν η περίπτωση της τουρκίας τα σύνορα με την οποία εξακολουθούν να αποτελούν την βασική είσοδο λαθρομεταναστών που ολοένα αυξάνει είναι ενδεικτική έχουν γίνει βήματα προόδου. ωστόσο η υπογραφή και η εφαρμογή συμφωνίας επανεισδοχής ευρωπαϊκής ένωσης τουρκίας είναι επιτακτική σήμερα όσο ποτέ. ανάλογη σημασίας είναι και η εφαρμογή της συμφωνίας ευρωπαϊκής ένωσης πακιστάν. στις περιπτώσεις της αλγερίας και του μαρόκο θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις όπως επίσης να ξεκινήσουν ανάλογες διαδικασίες με άλλες χώρες λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες λαθρομεταναστευτικές πιέσεις όπως οι βόρειες χώρες της, αφρικής η αίγυπτος το αφγανιστάν επίσης το ιράκ. Όσον αφορά τώρα τον έλεγχο του οργανισμού και μιας και το θέμα της διακοινοβουλευτικής αυτής σύσκεψης είναι η δημοκρατική λογοδοσία, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση η αναβάθμιση του στάτους του frontex σε ευρωπαϊκό οργανισμό ανάλογο της europol είναι μείζωνος σημασίας. δεν αφορά μόνο στην αποτελεσματικότητά του αλλά και στο δημοκρατικό κύρος της ευρωπαϊκής ένωσης. ο frontex πρέπει να αποκτήσει ενιαία και αμυγή ευρωπαϊκή υπόσταση. η στενή διασύνδεση και συνεργασία του frontex κυρίως με την europol καθώς και η αποστολή και οι αρμοδιότητες του οργανισμού που μπορούν δυνητικά να επηρεάσουν ανθρώπινα δικαιώματα επιβάλλουν τον δημοκρατικό έλεγχο της λειτουργίας του σαν ευρωπαϊκός οργανισμός θα υπόκειται πλέον στο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου όπως αρμόζει στα όργανα που διαχειρίζονται ανάλογα ζητήματα. γιατί είναι σημαντικό όταν μιλάμε για διεύρυνση με ευρωπαϊκούς όρους να μην λησμονούμε την διεύρυνση σε βάθος σε βάρος της διεύρυνσης σε πλάτος. η μέχρι τώρα αστοχία δημιουργίας θεσμικών αρμών εμβάθυνσης στις δημοκρατικές οι ρίζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει υπό αμφισβήτηση τη δημοκρατικότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Τα εθνικά κοινοβούλια λοιπόν οφείλουν να αναλάβουν ένα αυτόνομο πεδίο δράσης που θα προσβλέπει μια, μια διεκδίκηση, μια διεκδίκηση δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Frontex θα πρέπει να περνά και αυτός μέσα από αυτό το φίλτρο. Είναι γεγονός ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι η ευνοϊκότερη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όμως λυπηρή η διαπίστωση ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι δύο θεσμοί στους οποίους πετύχαμε την μεγαλύτερη πρόοδο βρίσκονται σε κρίση. Η Ευρωζώνη και η συνθήκη του Σέγγεν συνιστούν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ένωσης τους βασικούς πυλώνες ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. κι όμως εμείς οι ευρωπαίοι επιτρέπουμε πολλές φορές να τίθενται ανοιχτά υπό αμφισβήτηση. ο διάλογος που έχει ανοίξει περί μηχανισμών αναστολής της συμμετοχής σε συγκεκριμένους τομείς και επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταλλάσσουν το οικοδόμημα του κεκτημένου του σέγγεν η λύση δεν θα πρέπει να αναζητηθεί στον περιορισμό του κεκτημένου. αυτό θα αποτελέσει σαφή οπισθοδρόμηση στην πορεία για την ολοκλήρωση. αντιθέτως θα πρέπει να αναζητηθεί στην περαιτέρω ενίσχυση της έμπρακτης εφαρμογής αρχής αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. τις αρχές αυτές επιβεβαιώνει και η συνθήκη της λισαβόνας και θα ήταν πράγματι θλιβερό να τις αθετήσουμε δύο, μεγάλ... χρόνια μετά την υιοθέτησή Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση που αποκλίνει από τις αρχές της συνθήκες της Λισαβόνας μόνο βλαπτικά και διαλυτικά φαινόμενα μπορεί να προκαλέσει και να λειτουργήσει σε βάρος των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της Ένωσης και των πολιτών της. Αν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αναρωτιόμαστε τι τελικά θέλουμε, λιγότερη ή περισσότερη Ευρώπη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καλύτερα να αναλογιστούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν πληρώσει αρκετά θέλουν επιμένουν και ελπίζουν να μην χάσουμε αυτό το στίχημα. σας ευχαριστώ πολύ. Δεν αμφιβάλλουμε ότι ε, υπάρχουν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα και αντιμετώπισε και στο παρελθόν και ε, παρουσιάστηκαν πολύ καλά. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Τόμας Ρούλε από την Τσεχία για δύο λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τη θέση της τσεχικής γερουσίας σχετικά με την ε, θέση της Frontex, διότι υπερασπίζουμε ε, την ε, κατάσταση των ε, συνοριακών σταθμών και των κρατών μελών ε, πρέπει να στηρίξουμε τις ε, τις δραστηριότητες των κρατών μελών μέσω των οργανισμών αλλά δεν θέλουμε, είμαστε αντίθετοι στην ενίσχυση της θέσεως της Frontex για των συνοριακών αστυνομιών διότι πιστεύουμε ότι η Frontex ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό θα ήθελα να υποφεληθώ τις ευκαιρίες για να σας πω ότι η Frontex θα έπρεπε να συντονίζει και να επιμορφώνει. Δεύτερον, σχετικά με την προστασία των συνόρων. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στα εξωτερικά σύνορα, διότι τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ιδιαιτέρως είναι πολύ ευάλωτα, αλλά και τα ανατολικά σύνορα είναι εξίσου σημαντικά. Και θέλω τώρα να κάνω μία ερώτηση στην Ελίδα Ελληνίδα συνάδελφό μας. Μπορείτε να αξιολογήσετε ε, το πιλωτικό πρόγραμμα ταχείας επεμβάσεως στην Ελλάδα και θα ήθελα επιπλέον ε, αν έχω χρόνο να αναφερθώ στη χθεσινή συνεδρίαση για τον έλεγχο των ε, ευρωπαϊκών οργανισμών, τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αντιλαμβάνομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί είναι στενά συνδεδεμένοι αλλά κατόπιν της χθεσινής συζητήσεως έχω λίγο το συνέστημα και εδώ υπερβάλλω ότι υποβαθμίζονται τα εθνικά κοινοβούλια και απλώς θα ελέγχουν στα πλαίσια του συγκεκριμένου κράτους μέλους εάν ακολουθούν τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ το συζητήσουμε το θέμα αυτό αλλά στην τελευταία συνεδρίαση και τώρα η κυρία Μόνικα Λαμπέρτο Ευχαριστώ Κυρίες και κύριοι Ήμουνα αρχάρια πολιτικός και μία φίλη μου πολύ σοφή μου επέστησε την προσοχή στο ότι το θέμα του πότε κινείσαι είναι πολύ πιο σημαντική ίσως και από την κίνηση. Άρα η χρονικά επίκαιρη στιγμή είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό έχει αποδειχθεί. Όσον αφορά τη Frontex και την ασφάλεια γενικώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα για να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να επεμβαίνει κανείς την κατάλληλη στιγμή διότι ας θυμηθούμε την, ε, τις βόμβες στη Μαδρίτη, την επίθεση των τρομοκρατών που είχαν πολύ βαρύ τίμημα. Ήμουν τότε στην Ουγγαρία υπουργό και τότε ε, οργανώθηκε ε, μία έκτακτη συνεδρίαση στο Υπουργείο Εσωτερικών και διατυπώσαμε προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια στην Ευρώπη μέσω και ανταλλαγής ε, πληροφοριών και συνεργασίας των αστυνομικών και εφαρμοστικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι τα γεγονότα μας υποχρέωσαν αλλά η Frontex ήδη το 2008 είχε ζητήσει να ε, διευρυνθεί το νομικό της πλαίσιο άρχισαν οι διαπραγματεύσεις και φέτος στην Λιβύη ε, και στα νότια σύνορα άρχισαν οι επαναστάσεις ε, και γι' αυτό ε, τα γεγονότα βλέπετε ότι μας υποχρεώνουν να επιταχύνουμε τη λήψη των αποφάσεων. Τώρα όσον αφορά τη δημοκρατική εποπτεία του Κοινοβουλίου και τη την εξέταση για νομιμότητα και ε, ε, τα δικαιώματα ε, του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό πρέπει να επιβραδύνει την ταχύτητα λήψεως αποφάσεων διότι υπάρχουν ραγδαία γεγονότα τα οποία διαμορφώνονται διεθνώς και εμείς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ανα πάσα στιγμή γι' αυτό και σας λέγω ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις και νέες απειλές γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες της Frontex ε, ιδίω όσον αφορά τους ελέγχους στα σύνορα και εδώ διαφωνώ με τον Τσέχο συνάδελφο διότι πιστεύω ότι και οι ευρωβουλευτές και οι εθνικοί βουλευτές φέρουν μεγάλη ευθύνη επί του θέματος. Ο Γενικός Διευθυντής της Frontex είπε ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις, απλώς εφαρμόζει τις αποφάσεις και αυτό είναι σωστό αλλά η σημασία των ελέγχων δεν, δεν είναι λόγος για να επιβραδύνουμε τη λήψη των, αποφάσεων Ο κύριος Αγκουράκης έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Frontex ε, είναι βασικό στοιχείο των μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της, ε, κατασταλτικής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους μετανάστες που υπεραλιστικές επεμβάσεις όπως είναι αυτές του Αφγανιστάν ή της Λιβύης τους αναγκάζουν να επιχειρήσουν να επιβιώσουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα αυτά όμως στοχεύουν και τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζοντας στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα προωθούνται εξελιγμένοι μηχανισμοί παρακολούθησης και ηλεκτρονικού φακελώματος αξιοποιώντας βιομετρικά δεδομένα δορυφόρου κατασκοπευτικά αεροσκάφη γιγάντωση των δυνάμεων συνοριοφυλακής και στρατιωτικοποίηση στα πλαίσια του frontex. η πολιτική αυτή προκρίνει την ανάπτυξη μεγάλων δυνάμεων που θα κλείνουν τα σύνορα και θα αφήνουν στο όλιο των δουλεμπόρων του εξαθλιωμένους μετανάστες με σχεδόν βέβαιη κατάληξη των θάνατό τους είναι πάρα πολλά τα γεγονότα και τα συμβάντα με χιλιάδες πληγμένους στη Μεσόγειο, ε, γεγονότα που θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο και λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, αλλά και της αστάθειας, αλλά και λόγω της καπιταλιστικής παγκόσμιας κρίσης. Στοιχείο της ίδιας πολιτικής είναι να στηβάζουν τους μετανάστες σε άθλιες συνθήκες σε διάφορα στρατόπεδα και στη συνέχεια να τους προωθούν με τη βία στις χώρες καταγωγής όπου θα βρίσκονται αντιμέτωποι ξανά με τεράστιους κινδύνους για τη ζωή τους. Χαρακτηριστικό για την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η οδηγία για την επαναπροώθηση των μεταναστών που προβλέπει κράτηση μέχρι και 18 μήνες, απέλαση και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πενταετία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Σύμφωνο Δουβλίνο 2 με τα τρομακτικά προβλήματα που δημιουργεί σε εκατοντάδες χιλιάδες εγκλωβισμένους σε άθλιες συνθήκες μετανάστες στην Ελλάδα. Είναι προφανέ για μα ότι τα προβλήματα δεν πρόκειται να τα λύσει ούτε ο Frontex, ούτε η καπιταλιστική ανάπτυξη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει μια πολιτική ενάντια στου μετανάστε ώστε να του έχει φτηνή εργατική δύναμη. Γι' αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε για νομοποίηση όλων των μεταναστών, κατάργηση του Δουβλίνου 2, εξασφάλιση ίσων εργασιακών κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε περίθαλψη, υγειονομική φροντίδα, εκπαίδευση και κοινωνικέ παροχέ. Αγωνιζόμαστε να μπει ένα τέρμα στην κατασταλτική πολιτική, να διαλυθεί ο Frontex όπω πρέπει να διαλυθεί και το λαϊκό οικοδόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ κύριος Μάικλ Φελτσόν από το Κοινοβούλιο της Μάλτας. Ευχαριστώ. Προέρχομαι από το μικρό νησί της Μάλτας και ξέρετε ότι γεωγραφικά βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον προέρχομαι από εκεί, μάλλον είναι αναμενόμενο ότι θα μιλήσω για το θέμα αυτό. Ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στο ρόλο της Frontex και στο ρόλο της σε σχέση με την λαθρομετανάστευση ή την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως είπε ο κ. Λέτινεν στην παρουσίασή του. Εμείς ε, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε όσα βιώνουν οι Έλληνες ε, συνάδελφοι. Θέλουμε ε, περαιτέρω ενδυνάμωση και εξέλιξη του ρόλου της Frontex και πάλι θέλω να αναφερθώ στο θέμα της μεταναστευτικής διαχείρισης. Και αναφέρθηκε και το θέμα από τους συναδέλφους των επιχειρήσεων επιστροφών των μεταναστών. Έχοντας κατά νου την κατάσταση που ισχύει στη Μεσόγειο, ίσως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αποσαφινιστεί περισσότερο, δηλαδή να ε, το έχουμε κατά νου όταν εξετάζουμε εκ νέου και να διατυπώνουμε τους κανόνες περί Frontex στο παρελθόν. Η χώρα μου έχει συμμετάσχει και έχει φιλοξενήσει και επιχειρήσεις Frontex. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο τα τελευταία δύο έτη και μπορώ να σας πω ότι η χώρα μου ε, αποφάσισε να μην ε, φιλοξενήσει τη Frontex επειδή άλλαξαν ε, οι κανόνες επιχειρησιακοί της Frontex. Ίσως αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αποσαφινιστεί κυρίως όταν ακούμε εδώ τόσα πολλά λόγια για την Ευρωπαϊκή Ελληνική, τον επιμερισμό του βάρους κτλ. Και τα τελευταία χρόνια η Frontex ήταν πολύ πιο ενεργή στα ελληνοτουρκικά σύνορα και αυτό είναι κάτι που το έθιξε και η Ελληνίδα συνάδελφος. Ε, αναφερθήκατε και στο Δουβλίνο 2. Ίσως δεν είναι άμεσο θέμα συζήτησης εδώ, αλλά είναι σχετικό. Και θα ήθελα να πω κάτι, θα προσπαθήσω να σεβαστώ και το χρόνο. Αυτός ο οργανισμός έχει διαδραματίσει ένα ρόλο για ε, την νόμιμη μετανάστευση, όποια κριτική και αν έχει γίνει, έχει διαδραματίσει ένα ρόλο προς τη μία προ την άλλη κατεύθυνση. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να δούμε και ποιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει ε, σε σχέση με το τι γίνεται στις χώρες ε, της Βόρειας Αφρικής και το τι θα επακολουθήσει κατόπιν των εξελίξεων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ρότζερ Χέντεγα από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Για τις εξηγήσεις σας για το Frontex. Είναι επίκαιρο θέμα στο Σουηδικό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ και τον κύριο Μπουσουτήλ που μας μίλησε για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τον τρόπο επιτήρηση εποπτείας της λειτουργίας του Frontex. Έχω όμως ένα ερώτημα προς τον Διευθυντή Λάιτεν. Μίλησε για δυνατότητες που υπάρχουν να βελτιωθεί η λειτουργία και η καθημερινή ζωή στα κράτη-μέλη και συμφωνούμε, αλλά ταυτόχρονα μερικά κράτη-μέλη επικρίνουν το Frontex λέγοντας ότι πρέπει να κάνει περισσότερες προσπάθειες να είναι πιο αυστηρό και ο μηχανισμός εποπτείας του Σέγγεν απαιτεί την εφαρμογή ορισμένων κριτηρίων. Γι' αυτό, γι αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Γι' αυτό ερωτώ. Κύριε Λάιτενεν, βλέπετε κανέναν φραγμό, νομικό φραγμό στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς σας γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς τους κοινοβουλευτικούς και κάτι άλλο που ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Είναι συμβατά όλα αυτά τα μέτρα που πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με με ό,τι άλλο έχει προαποφασιστεί. Θέλω να κάνω τέσσερα σχόλια. Καταρχήν, ένα πολιτικού χαρακτήρα σχόλιο. Ήρθα στο Ηνωμένο Βασίλειο ω μετανάστης ε, πρώτη γενιά. Γεννήθηκα στην Εμένη, η μου ήταν από την Ινδία. Θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη δεν είναι προορισμός νόμιμης μετανάστευσης. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας από τη λαθρομετανάστευση, δηλαδή από όσου ε, ε, εκμεταλλεύονται ανθρώπους που καταβαλούν πολλά χρήματα προκειμένου να έρθουν και να ζήσουν κατά κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ε, στους συνάδελφους από την Ελλάδα και παροτρύνω όλους τους αδελφούς να πάνε να επισκεφτούν την παραμεθόριο μεταξύ Τουρκίας και ε, Ελλάδας ε, εγώ ξέρω ότι ε, όλοι παραδέχονται ακόμη και Έλληνες βουλευτές ότι είναι κακή η κατάσταση εκεί αλλά το θέμα είναι ότι το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει μια κρίση έχουμε τεράστιο αριθμό εισερχομένων ανθρώπων και τελικά πολλοί από τους μετανάστες αυτούς θα καταλήξουν στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ ή σε οποιαδήποτε από τις χώρες μας γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει επιμερισμό του άχθους δηλαδή πρέπει να δώσουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη σε αυτές τις χώρε στα σύνορα. Σε ό,τι αφορά τη Frontex, εγώ υποστηρίζω, η Επιτροπή μου υποστηρίζει το δουλειά τη Frontex, αλλά πιστεύω ότι από επιχειρησιακή σκοπιά θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο ρόλο για τη Frontex. Θα πρέπει να τη δοθεί η ικανότητα να αντιμετωπίσει ορισμένα από αυτά τα ζητήματα και όχι απλώ το νομικό πλαίσιο. Η επιτυχία τη Frontex στα ελληνοτουρκικά σύνορα έγινε μέσω ε, των ομάδων Rabbit. Ε, είχαμε ε, από τις 132.000 ε, μείωσε στις 43.000 στις εισρωές των μεταναστών και νομίζω ότι διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο η Frontex εκεί με τις επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρχει και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών Frontex, Europol, όλοι αυτοί οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί πρέπει να συνεργαστούν. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έκλεισα τον καταλογό των ομιλητών, αλλά έχουμε τέσσερις ακόμη που ζητούν το λόγο και αν σεβαστούμε το χρόνο θα έχουν με λιγότερο χρόνο οι ομιλητές από το πάνελ για να απαντήσουν. Περίπου ένα τέταρτο. Κύριε Πάντζο από την Τσεχία, το Τσεχικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για το Διευθυντή της Frontex. Αφορά τα εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία. Να σας πω ότι το σχέδιο Σέγγεν ε, αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για την τσεχική δημοκρατία, δηλαδή μας επέτρεψε την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ορισμένα προβλήματα ε, και έτσι ξεκινά μια συζήτηση σε σχέση με τις αρχές ε, Σέγγεν. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση για τη βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Δεν θα είναι ε, πλέον απαραίτητο να έχουμε ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα που δυστυχώς τα τελευταία, τελευταία έχουμε δει να εφαρμόζουν κάποια κράτη ο ρόλο της Frontex θα πρέπει να μείνει σε επίπεδο συντονισμού, υποστήριξη των δραστηριοτήτων των κρατών μελών στα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει την απόφαση ο Frontex να έχει και τα δικά του μέσα, να έχει τη δυνατότητα να προσλευει συνοροφυλακε συνοροφύλακες από άλλα κράτη-μέλη. Αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, αν ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σήμερα Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πρόσθετος λόγος ε, να μην κλείνουμε τα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην επανεντάσουμε δηλαδή τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Σε ό,τι αφορά την τσεχική δημοκρατία, να σας πω ότι είχαμε προβλήματα στα ε, σύνορά μας με τη Γερμανία. Εμείς ε, θέλουμε στο ε, μέλων ε, να γίνεται σεβαστή και δική μας πρακτική έλεγχου στα σύνορα. Επίσης ε, θεωρούμε ότι αν πρέπει για έκτακτους λόγους να επανεισαγάγουμε τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο εάν ε, υπάρχουν ε, απειλές ε, κατά της δημοσίας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας. Το να διευρύνονται οι λόγοι αυτοί, δηλαδή να καλύπτεται και η μετανάστευση, εγώ θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάχρηση αυτού του μέσου, αυτού του εργαλείου. Τώρα, ερώτησή μου στον κύριο Λαϊτίναν, τι πιστεύετε ως ε, προς την ε, θέσπιση ελέγχων για λόγους ε, κακοδιαχείρισης μεταναστευτικών ροών. Πιστεύετε, ε, όπως και εγώ, ότι αφού έχουμε ενισχύσει την έλεγχο στο εξωτερικά σύνορα, δεν χρειαζόμαστε πλέον τόσο να προστατεύσουμε τα σύνορά μας στο εσωτερικό του χώρου Σέγγεν. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Κύριος Κάλβιν Χόκκινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω διαφορετική άποψη από τον τελευταίο ομιλητή. Επισκεφτήκα τη Βαρσοβία ε, μαζί με άλλους συναδέλφους ε, και επισκεφτήκαμε τη Frontex και συζητήσαμε ναι, το πόσο δύσκολο είναι να ελέγξουμε την ελευθερομετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε γιατί να μην ε, έχουμε αυστηρούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για τους πολίτες τρίτων χωρών και θέτω αυτή την ερώτηση και πάλι σήμερα γιατί θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος έτσι ώστε να αναχαιτήσουμε και τους εγκληματίες και τους ελευθερομετανάστες. Η στα εσωτερικά σύνορα. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι όταν ε, περάσουν από τα εξωτερικά σύνορα μπορούν πολύ εύκολα να περάσουν τα εσωτερικά σύνορα. Ενώ αν έχουμε ελέγχου ε, στα διαβατήρια δεν θα είναι ε, τόσο εύκολο. Κάποιου μήνε αναφέρθηκε στο Βρετανικό τύπο ότι κάποια κράτη-μέλη ανησυχούσαν για τη Σέγγεν για ακριβώ τέτοιου λόγου και μάλιστα ένα κράτο μέλο είχε σκεφτεί να επανεισαγάγει τους ε, ελέγχους στα διαβατήρια ε, ακριβώς για αυτούς τους λόγους εμείς δεν είμαστε μέλος ε, του χώρου Σέγγεν και ούτε πρόκειται να γίνουμε γιατί η κυβέρνησή μας ε, θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο στα σύνορά μας. Εγώ προτείνω ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη στη Μεσόγειο καθώς οι λαθρομετανάστες θα ξέρουν στη συνέχεια ότι δεν μπορούν να διασχίσουν ε, και να περάσουν στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεώθηκε χτες ότι η έλεγχη Σέγγεν και άλλοι συνορική έλεγχη είναι θέμα συνεργασία και όχι εναρμόνισης Δεν είναι ομοσπονδιακή δομή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, οι διευθετήσει για τα σύνορα απαιτούν μια διαρθρωτική συνεργασία. Εγώ είμαι σίγουρο ότι οι περισσότεροι Βρετανοί, όπω ε, και εγώ, ε, θεωρούν ότι πρέπει να περιορίσουμε αυτή την κυκλοφορία. Ευχαριστώ κύριο Αντρέγη Χάνκο από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αγκουράκης μπορώ να συμφωνήσω μαζί του διότι πέρυσι είχα την ευκαιρία εδώ να παρουσιάσω τις ε, κριτικές των ανθρωπιστικών οργανώσεων έναντι της Frontex αλλά ε, ακόμη και πριν από λίγες εβδομάδες ε, το Human Rights Watch είπε πόσο βρώμικα είναι τα χέρια χέρια της Frontex σχετικά με ε, την αντιμετώπιση των κρατουμένων στην Ελλάδα και πρόκειται ε, για ε, λαθρομετανάστες. Βλέπουμε ότι αυτούς τους συλλαμβάνει η Frontex και τους έχουν σε απαράδεκτες συνθήκες να κρατούνται στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτές οι συνθήκες κρατήσεως είναι υποβιβαστικές για τον άνθρωπο και άρα η Frontex δεν εφαρμόζει τις ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές και αυτό το έχει πει ο Bill Frontley του Human Watch και λέγει ότι ακριβώς τη στιγμή όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει λάβει μία σημαντική ε, απόφαση ότι η ε, μεταφορά των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βλέπουμε τι συμβαίνει και να μία ερώτηση εις ε, την Ελλάδα και την Τουρκία γιατί ε, στα σύνορά τους ε, κατασκευάζεται ένα χαντάκι και από τη μία πλευρά θα υπάρχουν τάγκς από πλευρά της Τουρκίας και από την άλλη πλευρά θα έχει λάβει και η Ελλάδα μέτρα θα ήθελα να ξέρω εάν η Frontex Frontex συμμετέχει ή πρόκειται για μια ανεξάρτητη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Επίσης, όσον αφορά το οικοδόμημα της Frontex, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν μπορεί ο οργανισμός αυτός να τα αποτρέψει. Δηλαδή, ε, τι ε, αρμοδιότητες έχει και κατά πόσο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και επί της ουσίας. Η Τινησία έχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει τώρα διότι υπάρχουν 900.000 πρόσφυγες από τη Λιβύη. Δεν είναι σε θέση να το αντέξει και η Ελληνίδα συνάδελφος είπε ότι 132.000 πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα και φαντάζομαι ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κανείς να υποδεχτεί όλους αυτούς αρκετά αξιοπρεπώς ε, και κατακρίνω και την ε, γερμανική κυβέρνηση για τη στάση της. Πώς μπορεί όμως ε, να το αντιμετωπίσει την Ισία και δεν μπορεί η Ευρώπη διότι μιλάμε για αλληλεγγύη. Δεν χρειάζεται αλληλεγγύη μόνο για να αποφεύγουμε τους πρόσφυγες γιατί ουσιαστικά οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι εγκληματίες, είναι σε άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια έκτακτη κατάσταση. Ευχαριστώ και ο κύριος Γκίντερ Κέσελ τώρα από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, Εγώ αντιμετωπίζω το θέμα αυτό από μια διαφορετική οπτική γωνία γιατί πιστεύω ότι η Frontex είναι μια επιτυχημένη ιστορία και ε, μπορεί να συμβάλλει εις την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πράγμα που πρέπει να απασχολεί όλους τους Ευρωπαίους γι' αυτό και θεωρώ ότι η αναβάθμιση της Frontex είναι ποιοτικά πάρα πολύ σημαντική για να έχουμε μία αναβάθμιση και της προστασίας των συνόρων ε, και για να μπορούν να ελέγχονται και ε, οι διερχόμενοι ε, και η Ελλάδα μας είπε πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του οργανισμού αυτού στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Άρα θέλω να ρωτήσω τι υπάρχουν, τι είναι οι δυνατότητες και τι χρειάζεται η Frontex ακόμη για να μπορέσει να εξυπηρετήσει και να στηρίξει καλύτερα τις ε, εθνικές ε, ε, αρχές. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διότι εκφράστηκαν πάρα πολλές απόψεις που είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνεται όταν ε, ε, συγκεντρώνονται και ε, συναλλάσσονται τα 7 ευρωπαϊκά, τα 27 εθνικά κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τη Frontex όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε είμαστε ε, πιο επικριτικοί και γι' αυτό οργανώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Θα δώσω τώρα πρώτα τον λόγο στον κύριο Λάιτεν και μετά στα άλλα δύο μέλη ε, του προ... Ε, της Τράπεζας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν εδώ τις απόψεις τους και τις ερωτήσει. Θα απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις ε, διερώντας σε τέσσερα μέρη και στο τέλος ε, θα φτάσω και στην ερώτηση του Αυστριακού συναδέλφου. Καταρχήν, να αναφερθώ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως είπε ο κ. Μπουσουτήλ. Είναι ήδη αρκετά πλήρης και πρόσθετα έχουμε και κάποιους άλλους ε, πολιτικούς ε, οργανισμούς, κάποια άλλα πολιτικά όργανα, όπως η Κομισιόν και το Συμβούλιο, διαδραματίζουν ε, το ρόλο τους ως συνομοθέτες ή ως δημοσιονομική αρχή. Και είδαμε ότι ο αντίκτυπος αυτών των, η επιρροή αυτών των ευρωπαϊκών θεσμών αυξάνεται ως προς τη Frontex. Έτσι λοιπόν ο δημοκρατικός έλεγχος είναι αποτελεσματικός. Και υπάρχει δυνατότητα επιχειρησιακής ανεξαρτησίας στο βαθμό που χρειάζεται. Τώρα, το δεύτερο σχολείο μου είναι το εξή. Θέλω να προσπαθήσω να πεικονίσω το ρόλο των κρατών μελών. Η συνθήκη της Λισαβόνας ρητά αναφέρει ότι οι αποφάσεις ε, λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη και ε, η ευθύνη των επιδόσεων έγκυται στα κράτη-μέλη. Η Frontex δεν θέλει να αφαιρέσει αυτές τις αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα σαφές σημείο αφετηρίας για οτιδήποτε κάνουμε και πρέπει να είναι κατανοητό. Πρέπει να γίνει κατανοητό με τον σωστό τρόπο. Η Frontex είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας των κρατών μελών. Αυτό βασιζόταν σε αιτήματα, γινόταν με κούσια βάση, αλλά τώρα θα λάβει ένα πιο υποχρεωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή να υπάρχει συντονισμός της Frontex για την για το υπηρεσιακό σκέλο ε, των ε, επιχειρήσεων. Ε, δηλαδή, εμείς δεν λαμβάνουμε αποφάσει εκ μέρου των κρατών μελών, απλώ είμαστε υπεύθυνοι για το συντονισμό. Το τρίτο σχόλιο μου είναι αρκετά ενδιαφέρον και σχετίζεται με το θέμα της διαχείρισης της μετανάστευσης και τη λατρομετανάστευση. Ο έλεγχος των συνόρων είναι το κλειδί για όλα τα προβλήματα. Πρέπει να το ξεχνάμε Πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Δεν ισχύει. Είναι ένα τμήμα της λύσης, αλλά δεν είναι η συνολική λύση. Τι είδαμε πρόσφατα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είδαμε είναι ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται τόσο με την ικανότητα για την έλεγχο και την εποπτεία των συνόρων υπάρχει ε, πραγματικά μια μειοψηφία ε, διελεύσεων ε, μη ανιχνεύσιμων στα σύνορα. Το πρόβλημα είναι οι επακόλουθες διαδικασίες. Και αναφέρθηκε αυτό εδώ, πώς η διαδικασία ασύλου, πώς το σύστημα ασύλου λειτουργεί, πώς ε, λειτουργεί το σύστημα επιστροφών ε, των ατόμων που έχουν συλληφθεί και δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην επικρατεία των κρατών μελών. Όταν ε, δεν λειτουργούν ε, αυτά τα δύο συστήματα όπως πρέπει, δεν μπορεί να βρεθεί λύση μέσω των ελέγχων στα σύνορα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μαζί. Και αυτές οι δύο διαδικασίες ε, που σχετίζονται με το άσυλο και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρόλων και των επιστροφών, αν δεν υποστηρίζονται από ένα αξιόπιστο σύστημα συνοριακού ελεγχού, δεν λειτουργούν. Όλα αυτά τα μέσα τα χρειαζόμαστε λοιπόν και κάτι ακόμη για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι ε, πραγματικά κάτι που ενσωματώνεται στην ίδρυση του οργανισμού, στις αξίες του οργανισμού. Είμαστε δεσμευμένοι, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα προάγουμε. Και έχουμε ε, ουσιαστικά πολλές δράσεις για το πώς προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια του συνοριακού ελέγχου. Έχουμε εγκρίνει τη στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το σχέδιο δράση. Ο τροποποιημένο κανονισμό μα δίνει περισσότερε δυνατότητε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Έχουμε και τον αξιωματικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα το αναφέρω και ο κύριος Μπουζετήλα, έχουμε τον κώδικα διοντολογίας, έχουμε την κατάρτιση που σχετίζεται με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης έχουμε τις εκθέσεις για ε, να καταγγέλλονται ε, κάποιες περιπτώσεις όταν υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επίσης ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι οι κριτικές είναι επικοδομητικές για το μέλλον. Ε, δείτε την έκθεση της ε, Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Σεβασμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η έκθεση αυτή μας έδειξε ότι η Frontex δεν ήταν τόσο δραστηρία σε σημεία όπου είχαμε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τώρα σε σχέση με το τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε δέσμευση, συμμετοχή των κρατών μελών, συνεισφορά των κρατών μελών ε, με ένα συνεπή τρόπο, εφαρμόζοντας κοινού κανόνες ε, για, την, ε, για το συντονισμό. Αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ας συνοψίσουμε τώρα. Το Frontex θεωρούμε ότι είναι τιμήμα της λύσης και όχι του προβλήματος. Λοιπόν, ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσους συμμετέσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Θα κάνω μερικά σχόλια. Πρώτον, τα εξωτερικά σύνορα είναι κοινή ανησυχία όλων. Μερικοί συνάδελφοι είπαν ότι τα εξωτερικά σύνορα είναι θέμα εθνικής δικαιοδοσίας και έχουν βέβαια δίκιο. Αλλά και όμως πρέπει να ανησυχούμε και για τα εξωτερικά σύνορα του Σέγγεν, ας πούμε η τσεχική δημοκρατία πρέπει να ασχολείται όχι μόνο με τα δικά της σύνορα αλλά και με τα εξωτερικά σύνορα του Σέγγεν. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσουμε και Φάνηκε πόσο σημαντικό είναι το ερώτημα αυτό φέτος όταν η Γαλλία χρειάστηκε να επαναφέρει τους ελέγχους στα εθνικά της σύνορα σε ένα σεγγενικό σύνορο, δηλαδή Γαλλίας-Ιταλίας. Και ο λόγος που το έκανε δεν ήταν επειδή υπήρχε πρόβλημα με το εσωτερικό αυτό σύνορο με την Ιταλία, αλλά λόγω των εξωτερικών σύνορων της Ιταλίας, δηλαδή το νησί της Λαμπεντούσας. Άρα εκείνοι που έλεγχαν τα σύνορα στη Λαμπεντούζα αν πίεσαν τη Γαλλία η οποία αναγκάστηκε να επαναφέρει ελέγχου στα δικά της σύνορα. Το μάθημα που παίρνουμε από αυτό είναι ότι τα εξωτερικά σύνορα της Λαμπεδούσης δεν είναι απλώς ιταλικό θέμα αλλά και γαλλικό και τσεχικό και του καθενός και της καθεμιάς. Δεύτερον, μήπως δημιουργούμε μία πανενοσιακή αστυνομία των συνόρων, όχι. Όχι, γιατί, όπως είπε και ο κύριος Λάιτεν, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν 400.000 υπεύθυνοι για τους ελέγχους στα σύνορα σε ολόκληρη την Ένωση και θα ήταν παρανοϊκό να πούμε ότι πρέπει να το, ξανα, να το πολλαπλασιάσουμε. Υπάρχουν ήδη αυτοί. Το θέμα είναι να υπάρξει μια υπηρεσία που να λειτουργεί, μάλλον να την κάνουμε πιο αποτελεσματική την υπηρεσία που υπάρχει, βασικά στα σημεία των εξωτερικών μας συνόρων που είναι τα πιο αδύνατα, τα πιο εκτεθειμένα, έτσι ώστε να είναι φανερό ότι τα εξωτερικά σύνορα είναι τόσο ισχυρά όσο ο αδυναμότερος τους κρίκος. Πρέπει λοιπόν να, είμα, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κάποια αξία στην ευρωπαϊκή συνεργασία και για το θέμα αυτό του ελέγχου των εξωτερικών σύνορων. Τρίτον, ο συνάδελφος από τη Μάλτα δικαίως ανέφερε τις κατευθυντήριες γραμμές που αλλάζουν τους κανόνες για την παρέμβαση του Σέγγεν. Όντως δεν είναι αυτό το τμήμα του κανονισμού του Frontex που πρόσφατα άλλαξε. Αλλά ε, το επηρεάζει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα της αλλαγής των κατευθυντηρίων γραμμών λειτουργίας του Frontex. Φέτος 50.000 περίπου άνθρωποι κατέφτασαν στη Λαμπεντούσα ενώ 1.500 στη Μάλτα, τη δική μου χώρα δηλαδή. Η Λαμπεδούσα και η Μάλτα απέχουν περίπου 150 χιλιόμετρα και η τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αριθμών αφήξεων μας δείχνει αμέσως ότι οι μετανάστες ήξεραν πού ακριβώς ήθελαν να πάνε. Ήξεραν ότι αν έφταναν στη Μάλτα θα... δεν θα μπορούσαν να ξαναφύγουν, ενώ στη Λαμπεντούσα οι Ιταλικές αρχές θα τους πήγαιναν στην Ιταλία, στο Ιταλική Ήπειρο. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτό η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δηλαδή να αναλάβει η Μάλτα το πρόβλημα της Λαμπεντούσας και τα λοιπά. Και γι' αυτό αρνήθηκε τη συμμετοχή της στο Frontex, πράγμα το οποίο είναι βέβαια τραγική ηρωνία γιατί όντως η Μάλτα χρειάζεται παραπάνω από άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα και η Ιταλία βέβαια το Frontex γιατί εκτίθεται ιδιαίτερα πολύ. Τέλος, η κατάσταση στην Τινησία. Κάποιος είπε ότι πολλοί έφυγαν από τη Λιβύη για να πάνε στην Τινησία. Πράγματι, 3 τέταρτα πενήντα περίπου. Από αυτούς, πολλοί επέστρεψαν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως, που έστειλαν πτήσεις από τα σύνορα της Τινησίας προς διάφορες χώρες από που προέρχονταν αυτοί οι πρόσφυγες. Αλλά 60.000 περίπου Λίβοι παρέμειναν στην Τινησία και μένουν με οικογένειες εκεί. Και περίπου 4.000 μένουν εκεί στην έρημο στα σύνορα μεταξύ Τινησίας και Λιβύης. Και αυτοί μένουν εκεί σε συνθήκες ερήμου γιατί δεν έχουν που να πάνε. Υπάρχουν χώρες όπως η Σομαλία, η Ερυθρέα, το Σουδάν είναι από την Ερυθρέα, τη Σομαλία και το Σουδάν και δεν μπορούμε να τους ξαναστείλουμε εκεί. Πράγμα το οποίο θέτει το ερώτημα εάν η, Τουνησία, η Τινησία εκφράζει τέτοια αλληλεγγύη για 750.000 ανθρώπους δεν θα έπρεπε και ο ανεπτυγμένος κόσμος να επιδείξει ανάλογη αλληλεγγύη για τις τέσσερις αυτές χιλιάδες που μένουν εκεί στην έρημο. Οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν αποτελέσει υπόδειγμα. Είπαν εγώ αναλαμβάνω όσο το δυνατόν περισσότερους και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έπραξε κάτι ανάλογο. Αν δεν αντιδράσουμε λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να έρχονται στην Ευρώπη με παλιόβαρκες και θα, κινδυνεύουν, θα διακινδυνεύουν τη ζωή τους και γενικώ θα διαβιούν με αναξιοπρεπή τρόπο. Υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα βέβαια για αυτούς που είναι στα σύνορα με την Τινησία. Το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο της Λιβύης ελέγχει αυτή τη στιγμή τα πράγματα και μπορούν να επιστρέψουν είναι και αυτή μια δυνατότητα, αλλά όχι για αύριο βέβαια. κυρία Τσολόγλου. Ε, θα ήθελα και εγώ να συνοψίσω και να συμπυκνώσω τις διαπιστώσεις ε, των ε, συμμετεχόντων. θα πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι η Ελλάδα έχει δεχτεί ένα απίστευτο κύμα μεταναστευτικών ροών κατά την τελευταία πενταετία αυτό σημαίνει ότι δέχτηκε τέτοιες συνθήκες όπου δεν μπορούσε να τις είχε προνοήσει γιατί αυτά δεν εξαρτώνταν από τη δική της βούληση και τη δική της ε, πολιτική ιδίως από περιοχές ε, της τουρκίας ε, όπου συσσωρεύονταν πακιστανοί αφγανοί και λοιποί όπως επίσης και από τις βόρειες χώρες της αφρικής και βέβαια δεν είχε την απαραίτητη υποδομή και τις δυνατότητες και τα εργαλεία ώστε να ανταποκριθεί ε, και να οργανωθεί ακέραια και άριστα ε, μια υποδοχή αυτών των παράνομων μεταναστών ε, και βεβαίως δεν μπορεί να την αδικεί την χώρα μου το γεγονός ότι προσπάθησε άμεσα να ε, δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης όπου βελτιώνονται οι συνθήκες παροχής ασύλου όπου ε, βελτιώνονται ε, και εξετάζονται οι αιτήσει αυτών που πρέπει να τύχουν της διεθνούς προστασίας αλλά και να είναι αυστηροί σε όσους αναπτύσσουν παραβατικές συμπεριφορές. Ε, αξίζει να σας πω ότι το 70% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί και αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί πράγματι ε, εκείνοι οι οποίοι έρχονται στη χώρα δυστυχώς αναπτύσσουν και παραβατικές ε, συμπεριφορές. Ε, επίσης θέλω να τονίσω ότι το 80% των λαθρομεταναστών και χαίρομαι που αυτό το διεπίστωσε η πλειοψηφία των ομιλητών είναι λαθρομετανάστες οι οποίοι μέσω της χώρας μας διοχετεύονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. έρχονται και επιδίωξή τους είναι να φύγουν. γι' αυτό το λόγο και συσσωρεύονται στα δυτικά λιμάνια εκείνα που οδηγούν στην ιταλία όπως στην πάτρα και στην ιγουμενίτσα και με χίλιους τρόπους έστω και παράνομους παράνομους προσπαθούν να διαφύγουν. Αλλά έχει παρατηρηθεί ότι παρά την ε, ε, κινητοποίηση του Frontex, την βοήθεια του Frontex σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, ε, σε τεχνικό, προσωπικό και επιστημονικό, δυστυχώς ενώ μειώθηκαν οι εισρωές από τα θαλάσσια σύνορά μας, ε, και βεβαίως από τα χερσαία δεν έχουν μειωθεί από τα τουρκικά εκεί δηλαδή όπου είναι ο εύρος που είναι ένα φυσικό σύνορο και επειδή πλην του ποταμού αυτού δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια ώστε να κάνουν δύσκολη την πρόσβαση από τα βόρεια σύνορα προς την Ελλάδα αυτή ήταν και η ανάγκη που οδήγησε την χώρα μου, την κυβέρνηση ώστε να κατασκευάσει τον φράχτη αυτόν που λέμε μια τάφρο η οποία ε, περιφράσετε με σειρματόπλεγμα και βεβαίως να πολλαπλασιάσει τις επιχειρήσεις των «rabbits» του ακριβώ όπως ακριβώς επεσήμανε και ο φίλος ε, ο οποίος από ό,τι ε, κατάλαβα είναι μετανάστης από την Ινδία, ακριβώς για να παρεμποδίσει αυτήν την είσοδο την παράνομη. Δηλαδή, η είσοδος από την Τουρκία, ενώ στο προηγούμενο χρόνο ήταν γύρω στα 6.000 παράνομους μετανάστες, σήμερα έχει ξεπεράσει τις 9.000. Και αυτή τη στιγμή συνοστίζονται στα παράλια του Εύρου, του ποταμού αυτού που σας εξήγησα χιλιάδες ε, μετανάστες λάθρομετανάστες ε, οι οποίοι προέρχονται από χώρες τουρκία πακιστάν αφγανιστάν και άλλες χώρες της ανατολής περιμένουν να κατέβουν τα, ε, τα, του ποταμού τα νερά ώστε με πλαστικές βάρκες να εισέλθουν από τα σύνορα αυτά. είναι λοιπόν φυσικό επόμενο εφόσον είναι εθνική υπόθεση διαφύλαξη των ισόρων πρωτίστως να προσπαθήσουμε σαν κυβέρνηση να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας άρα αυτή η πράξη δεν είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμείς σαν χώρα οφείλουμε να ισορροπήσουμε αφενός μεν στο σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων προφανώς αλλά και στην διαφύλαξη της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας και του έθνους μας. με όλες αυτές λοιπόν τις ενέργειες και με τη συνεργασία με την frontex πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή ένωση αναγνωρίζοντας τον ότι ανατολικό άκρο της μεσογείου λόγω της γεωγραφικής του θέσης είναι και όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της, πιστεύουμε ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες αυτές αλληλεγγύης, οι προσπάθειες οι κοινέ ή επιχειρησιακές, αλλά και οι οικονομικές ενίσχυσης του Frontex, όπως επίσης τον ενισχύουμε και οι εθνικοί προϋπολογισμοί προφανώς, ακριβώς για να προστατευτεί η Ευρώπη από το κύμα των λαθρομεταναστών πιστεύω ότι είναι αυτή μια λύση δίκαιη και όλοι θα, πρέπει να, συνδράμουμε πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν οι απροσδόκητες εξελίξεις από την ε, βόρεια αφρική. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, ε, παρουσίασαν εδώ τις απόψεις τους και μας έκαναν σοφότερους ε, και μας ενημέρωσαν καλύτερα επί του θέματος. Ήταν πολύ ζωντανή συζήτηση και νομίζω ότι διασκέδασε τις ε, ιδέες ότι η Frontex δεν είναι μία σημαντική οργάνωση για μας και έφυξε και όλα τα οργανωτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον διευθυντή της Frontex για το ότι κάνουν και να συνεχίσουμε αυτό το έργο εποπτείας το οποίο ε, ξεκίνησε πολύ ζωντανά αυτή η συνεδρίαση να συνεχίσουμε δηλαδή για τα επόμενα έτη και θα ήθελα τώρα να κλείσω αυτή τη συνεδρίαση και να προσθέσω ίσως ε, ένα θέμα. Όπως ο κύριος Χόπκινς μας είπε, η χώρα μου δεν είναι πλήρες μέρος της ε, Frontex ε, όπως δεν είναι μέλος και του Σέγγεν αλλά ε, όταν η κυβέρνηση συνασπισμού δημοσίευσε τους στόχους της ανέφερε στη, την ενίσχυση της Frontex γιατί ακόμη και χωρίς να είναι μέλος του Σέγγεν αναγνωρίζει ότι η Frontex πρέπει να επιτύχει είναι δηλαδή μια σημαντική ένδειξη για το πόσο όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Και επειδή Έχουμε λιγότερο από δύο ώρες. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση σχετικά με το με ποιους τρόπους μπορεί τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσουν την κοινή του συνεργασία και εποπτεία των οργανισμών. Παρακαλώ λοιπόν τους υπευθύνους να έρθουν στο Προεδρείο και πρέπει να σας πω ότι ένας από τους ε, μιλητές ε, ε, δεν θα μπορέσει να έρθει. Πρόκειται για την κυρία Λάμπερτ και έχουμε τέσσερις ομιλητές αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές απόψεις οι οποίες θα παρουσιαστούν και μόλις ο κύριος Αγγιλάρ φτάσει στη θέση του ή θα καθίσει κάτω. θα ξεκινήσουμε με αυτόν σαν πρόεδρο της ε, συνεδριάσεως και όλης ε, της διοργανώσεως ε, και τον ευχαριστούμε για την εκδήλωση αυτή που οργάνωσε και ε, θα ξεκινήσουμε αλλά θέλω ακόμη να κάνω κάτι να σας πω ότι επί του θέματος είμαι εμπλεγμένος διότι η η Βουλή των Λόρδων έχει ε, δηλώσει, έχει δηλώσει ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και ε, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται ένας νέος οργανισμός να δημιουργηθεί. Είμαι σίγουρος ότι τώρα θα υπάρξει μία πολύ ζωντανή συζήτηση επί του θέματος αυτού και δίνω το λόγο στον κύριο Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Λόρντ Χάνι. Ε, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα εδώ να δώσω και εγώ την συνδρομή μου στο τελικό αυτό, στην τελική αυτή συνεδρίαση, συνοψίζοντας τη σημασία των βελτιώσεων τις οποίες ε, μπορούμε να επιφέρουμε ε, ε, μέσω της συνεργασίας την οποία έχουμε καταρτήσει ή στην αξιολόγηση της πολιτικής και ιδιαιτέρως ή στις επιδόσεις και εις ε, την ε, ε, απόδοση των οργανισμών αυτών που έχουμε καταρτήσει διότι αφού υιοθετήθηκε το πρόγραμμα το Δεκέμβριο του 2009 ξεκίνησε η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια Ξεκινήσαμε με την ε, ε, μόνιμη επιτροπή ε, επί της για θέματα εσωτερικής ασφαλείας, τη λεγόμενη κόζη και η στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας εγκρίθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2010 και περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για δράση. Δύο χρόνια όμως ε, μετά ε, ένα χρόνο μετά δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση και ε, χρειαζόμαστε ακόμη να καταρτήσουμε ε, την ε, κοινοβουλευτική εποπτεία και γι' αυτό συναντηθήκαμε διότι υπήρξε μία πρώτη κοινοβουλευτική συνεδρίαση τον Οκτώβριο του 2010 και τώρα θα έχουμε τακτικές συνεδριάσεις αξιολογήσεως για να παρακολουθούμε αυτές τις πολιτικές όπως άλλωστε και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την Europol, την Eurojust, τη Frontex, ε, όλες αυτές ε, εξετάστηκαν και παρουσιάστηκαν κατά το σεμινάριο αυτό των δύο ημερών και ε, πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία ήδη έχουν ληφθεί από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή α Επιτροπή, δηλαδή να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός κύκλος ο οποίος θα οριοθετεί την συνεργασία των ενδιαφερομένων από αυτό το χώρο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τονίσω αυτό το οποίο είπα και χθες μετά από την έναρξη της συζητήσεως, δηλαδή ότι είμαστε εδώ για να προσδώσουμε δώσουμε μία επιπρόσθετη αξία σε αυτές τις ρυθμίσεις, να βοηθήσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν για να βελτιώσουμε την ε, αξιολόγηση και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσουμε τις προτεραιότητες που έχουμε καταρτήσει ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εξωτερικά σύνολα, ε, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γι' αυτό ε, και εγώ ε, θέλω να τονίσω τη σημασία της συνεργασίας ε, να κάνουμε δηλαδή μία κοινή άσκηση και να καλέσουμε στα εθνικά κοινοβούλια ε, της, τους οργανισμούς αυτούς. Εμείς τους ε, ακούμε τακτικά, τους καλούμε στην Επιτροπή Ελευθεριών, παρουσιάζουν τις διάφορες, τα διάφορα θέματά τους, αλλά σύμφωνα με την νομική βάση που παρουσιάσαμε εχθες 70, 71, 86, 88 πρέπει να συνεργαστούμε τα ευρωπαϊκά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, για να γίνει σωστά η δουλειά και να υπάρχει ε, μία αντιπαραβολή των ε, ελέγχων οι οποίοι γίνονται και να αξιολογήσουμε την ε, απόδοση ε, των οργανισμών αυτών να αξιολογήσουμε την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν και κατά περίπτωση ε, να σκεφτούμε τι προσαρμογές χρειάζονται και από εθνικής και από ευρωπαϊκής πλευράς. Εάν γίνει κάτι τέτοιο στους επόμενους μήνες και προετοιμαστούμε να προβούμε εις αυτήν την προσαρμογή θα εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι συναντήσεις μας θα είναι όντως αποτελεσματικές για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ε, στους πολίτες και να τους ε, περάσουμε το μήνυμά μας. Δηλαδή, ε, εάν αυτές οι συνεδριάσεις είναι επιτυχείς, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ε, κάθε εθνικό κοινοβούλιο το οποίο θέλει ε, να συμβάλλει ε, στην αξιολόγηση αυτή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Νόσος σύμφωνα με το άρθρο 70 θα μπορέσει να επανέλθει και του χρόνου όταν στον Οκτώβριο του 2012 θα γίνει και πάλι αυτή η συνεδρίαση και ε, οι εθνικές εκθέσεις θα μπορέσουν να συμπληρώσουν τις παρουσιάσεις των οργανισμών και να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την ε, εθνική ε, προοπτική. Να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε διότι όλα αυτά πρέπει να συντελούνται σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτού ξεκινήσει η νέα διαδικασία μετά το 2013. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτές τις ε, πληροφορίες ε, μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια στα πλαίσια του ενιαίου χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας ε, με τις διάφορες επιτροπές οι οποίες εμπλέκονται και να διευρύνουμε τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε εις ε, τις ε, προσδοκίες των πολιτών από τις εφαρμογής αυτής ε, της νέας νομικής βάσης πέραν αυτού να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό το πληροφοριακό το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει επανειλημμένως διότι εδώ γνωρίζουμε ότι πολλές από τις πληροφορίες τις οποίες συγκεντρώνουμε έχουν άμεση ε, σχέση με τους οργανισμούς που εμπλέκονται δηλαδή το Europol, Eurojust, ε, τη Frontex και θα πρέπει ε, να, οι πληροφορίες αυτές να ενημερώνουν και σε εθνικό επίπεδο παντού τους πολίτες για να μπορούμε ε, να ε, βελτιώσουμε την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση αυτών των διαδικασιών. Έχουμε δηλαδή μια νέα λυσίδα η οποία θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή δημοκρατία και να αποτελέσει ένα προηγούμενο βάση του άρθρου 10 ε, των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε τώρα να ξεκινήσουμε, να θέσουμε σε κίνηση αυτή τη δυναμική, να προετοιμάσουμε την Δανική Προεδρία, να προετοιμάσουμε το επόμενο σεμινάριο του Οκτωβρίου 2012 και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε μία θετική απάντηση στις αιτιολογημένες αμφιβολίες οι οποίες ε, έχουν εκφραστεί για αυτές τις τακτικές συνεδριάσεις μας ε, και από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για να μην ε, είμαστε απλώς ικανοποιημένος, ικανοποιημένοι ότι εφαρμόζουμε τις επιταγές οι οποίες έχουν διατυπωθεί και ότι ε, σωστά ε, εφαρμόζονται όλες οι πολιτικές για τον χώρο ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλά. Νομίζω ότι καλό ήταν αυτό για την αρχή της ε, ε, συζητήσεώς μας και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πάολο Πίσκο, μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ζητήσω κατανόηση για το ότι θα πρέπει να φύγω νωρίτερα γιατί ε, έχω αεροπλάνο στις 12 και 20. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να παραβρεθώ εδώ και ε, να μπορέσω να σας παρουσιάσω την άποψη του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου για ένα θέμα που είναι τόσο σημαντικό για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα η δυνατότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων να μπορούν να παρακολουθήσουν θέματα που αφορούν εγγυήσεις, ελευθερίες και δικαιώματα αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την διαδικασία του, ε, του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος που ενισχύεται τώρα με τη Συνθήκη της Λισαβόνα και τη Χάρτα των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Οι Εθνικέ κοινέ γνώμες ε, πρέπει να γνωστέρουν ότι οι εκπρόσωποι τους προσδίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα όπως η περάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και τη σταθερότητα των κοινωνιών μα. Γι' αυτό είναι σημαντικό ε, η πολιτική, στη πολιτική μας ε, να εντάσσουμε την αποτελεσματικότητα με το σεβασμό των αξιών ε, του ευρωπαϊκού project όμως για να μπορεί η παρακολούθησή μας ε, να είναι αποτελεσματική έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Πολλές ε, από, πολλά από τα θέματα αυτά είναι ακόμα καινούργια στο ευρωπαϊκό ε, επίπεδο και επηρεάζει πάρα πολύ ο διακυβερνητικός χαρακτήρας των έλεγχο του. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν δεν πρέπει να είναι παθητικά, πρέπει να γνωρίζουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν αντιλαμβάνονται στους ε, τομείς που αφορούν ε, τις δραστηριότητες της COSI, της Europol, της Eurojust κτλ. Το άρθρο της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 61, αναφέρει ότι πρέπει τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, είναι ενημερωμένα από το Συμβούλιο για θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Ε, Όμω και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να παρακολουθούνται ευρύτερα. Ε, επίσης ε, φαίνεται να μην έχουν επαρκή γνώση τα κοινοβούλια σε σχέση με τις εργασίες αυτών των οργανισμών ασφαλείας και οι αρμοδιότητες, ε, μάλλον συγγνώμη, οι γνώσεις των Υπουργείων, των Οργανισμών Ασφαλείας και Πληροφοριών δεν αποτελούν πάντα προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι τα ευρωπαϊκά θέματα εξακολουθούν να παραμένουν κάπως απομακρυσμένα από τα ενδιαφέρον των εθνικών κοινοβουλίων. Έτσι λοιπόν η απάντηση που πρέπει να δώσουμε ε, είναι στην εξή ερώτηση. Με ποιο τρόπο μπορούν τα Εθνικά Κοινοβούλια να συζητήσουν αυτά τα θέματα στο ίδιο επίπεδο που συζητούνται και, στα, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια κυρίω θα επικεντρώνονται στα εσωτερικά θέματα, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, μάλλον ενώ τα ευρωπαϊκά ζητήματα θα παραμένουν ε, μη προτεραιότητα και πιο απομακρυσμένα. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε επαρκή έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τα εθνικά κοινοβουλία πρέπει να έχουν προδραστική ε, στάση και να προβλέπουμε συζητήσεις όπως είναι αυτή για να βελτιώσουμε, στην, ε, για να βελτιώσουμε τη λειτουργία των υφιστάμενων μηχανισμών. Ε, στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Πρέπει λοιπόν ε, να βελτιώσουμε το πώς ε, αντιλαμβάνονται τα Εθνικά Κοινοβουλία το έργο των οργανισμών, πώς συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές και πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Έτσι λοιπόν τα Εθνικά Κοινοβουλία θα πρέπει να αντελάσσουν εμπειρίες σε σχέση με το πώς γίνεται η παρακολούθηση υποπτία των θεμάτων αυτών. Όλες αυτές οι πτυχές είναι θεμελιώδες προκειμένου οι εθνικοί βουλευτές να μπορούν να παρεμβαίνουν με καλύτερο καλύτερο τρόπο σε τομεί. Τα εθνικά κοινοβούλια έτσι λοιπόν θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να κάνουν κριτική ανάλυση για τη λειτουργία των οργανισμών ασφαλείας που έχουν πάρα πολύ σημαντικό ε, ρόλο στην εκτίμηση της εγκληματικότητα, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην ανείχνευση των απειλών στην ασφάλεια. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν να συνεισφέρουν για τη βελτιότητα της αποτελεσματικότητά τους, για το σεβασμό των ελευθεριών των πολιτών και των δικαιωμάτων τους και για την παγίωση πολιτικών ε, και δράσεων που να συνάδουν ε, με τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν προσθεμένη αξία για μας του Ευρωπαίους η ενίσχυση του συντονισμού ε, της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ με τους ε, κυβερνητικούς οργανισμούς που υποπτεύουν των θεμάτων αυτών, κυρίως δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων, είναι κάτι πολύ σημαντικό για να έχουμε πιο αποτελεσματική εποπτεία. Νομίζω ότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που με τη συνθήκη της Λισαβόνας ρυθμίζεται ότι συμμετέχει σε όλα αυτά τα θέματα, μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο για την ανάλυση το πώς εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές, γιατί η εγκύτητά της στα θέματα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την εγκύτητα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όμως, εμ, παρά το ότι στέθηκε σε ισχύ σε συνθήκη, η συνθήκη της Λισαβόνας συνεχίζουν να υπάρχουν ε, πάρα πολλά διαφοροποιημένα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο και μπορεί να έχουν να κάνουν με διαφορετικούς ε, τρόπους καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος ή έλεγχο των συνόρων και έτσι λοιπόν ε, προκαλούν την εντύπωση ότι έχουμε ευρωπαϊκή απεικοδόμηση και έτσι λοιπόν ε, πρέπει να αποφύγουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή τα εθνικά κοινοβούλια ε, λίγα μπορούν να κάνουν ή τίποτα όταν ε, μιλάμε για την υιοθέτηση μέτρων που δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές συνθήκες και συμφωνίες όπως έγινε με την πρόσφατη επανεισαγωγή των ελέγχων στα σύνορα ε, που έγινε σε, μια, σε κάποια κράτη-μέλη ή όπως ε, αντιμετωπίστηκαν οι συνέπειες ε, της Αραβικής Άνοιξης. Πολλές φορές είδαμε ότι παραβιάστηκαν εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπήρχαν δυσκολίες να αντιμετωπιστούν τόσο δύσκολες καταστάσεις. Όμως τα γεγονότα αυτά ε, είχαν ε, ως ε, αποτέλεσμα να στρέψουν την προσοχή στη σύμβαση Σέγγεν και στη δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αναγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να προστατευτούν από τις απειλές στην εσωτερική ασφάλεια. Μάλιστα δεν πρέπει να διστάζουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία για να πετύχουμε με αποτελεσματικό τρόπο ε, το ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να αισθάνονται σίγουρα στο έδαφος τους. Ε, υπάρχουν ε, διάφορα μέτρη ε, γιατί ε, και έχουμε πάρα πολλές απειλές όπως ε, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα ακόμη και οι αναξέλεκτες μεταναστευτικές ροές. Αυτά τα φαινόμενα ποτέ δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα αν δεν υπάρχει καλή διάρθρωση μεταξύ των διάφορων ευρωπαϊκών και εθνικών οργανισμών με μια σοβαρή και εκδική παρακολούθηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα θέματα αυτά ε, θα πρέπει να τα προσεγγίζουμε πάντα έχοντας κατά νου τις ανθρωπιστικές αξίες τις οποίες θα πρέπει να τις υπερασπίζουμε κάθετα προκειμένου να εγγυθούμε το σεβασμό του κράτους δικαίου και της ελευθερίας των πολιτών και για το λόγο αυτό η συνεργασία των διάφορων οργανισμών με την υπηρεσία, με τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να είναι μόνιμου χαρακτήρα και απευθεία και να αποτελεί προτεραιότητα. Η αναγκαιότητα τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει σαφεί πολιτικέ που θα διευκολύνουν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι κάτι σημαντικό, ακόμα και αν γνωρίζουμε τι δυσκολίε που συνεχίζουν να υπάρχουν στο να συγκεράσουμε τι διάφορε οπτικέ ε, των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική πιο κοινή και καλύτερα διαρθρωμένη. Αυτό είναι απαραίτητο για να έχουμε πραγματική εποπτεία σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ο κύριος Κάρλος Κοέλιο μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο οποίος υπήρξε εισηγητής διαφόρων εκθέσεων για το κεκτημένο του Σένιγκεν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Αρχίζω από το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι πια αυτό που ήταν. Δεν είμαστε μόνο η Ευρώπη αγαθών και υπηρεσιών αλλά οικοδομούμε την Ευρώπη των πολιτών και έναν χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας. Όταν για πρώτη φορά αντιμετωπίσαμε την πρόκληση αυτή μετά τη σύνοδο του Τάμπερε αναζητούσαμε κυρίω καλύτερη και περισσότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Σήμερα όμω μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνας αναπτύσσουμε ευρωπαϊκά πραγματικά προγράμματα και κοινά πρότυπα νέου νόμου και εργαλεία. Οι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη εξέλιξη και η εντολή του και η δραστηριότητά τους μπορούν να συγκριθούν από αυτά που κάνουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες αλλά όμως χωρίς ομοσπονδιακό δημοκρατικό έλεγχο. Η θέση ενισχύ της συνθήκης Λισαβόνας ήταν το πρώτο βήμα για να δημιουργηθούν στενότεροι δεσμοί μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων με αποτέλεσμα πολύ καλύτερη συνεργασία αυτών των δύο τομέων. Οι δικαιοδοσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκείνες των Εθνικών για τον, προηγούμενο, για τον πρώην τρίτο πυλώνα συνεργασία για τη μετανάστευση και την αστυνόμευση έχουν αυξηθεί. Ιδιαίτερα από τότε που τέθηκε ενισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας που ενδυνάμωσε σαφώς τις δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου. Αλλά και όμως στην πράξη ακόμα πολλά πρέπει να γίνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται περισσότερο με τα εθνικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα δε εθνικά πρέπει να, έχουν να είναι πιο πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν τις νέες αυτές δικαιοδοσίες τους. Πρέπει να βρεθούν λύσεις για προβλήματα που δημιουργούνται από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να γνωμοδοτεί για τη σύναψη διεθνών συμβάσεων όπως για τα προσωπικά δεδομένα, χωρίς όμως καν να πληροφορούνται τα εθνικά. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη συνεργασία με τα εθνικά, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος, μονόδρομος είναι, για να υπάρξει δημοκρατική λογοδοσία. Ας δούμε τώρα τη λειτουργία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και των εντολών τους όπως η Ευρωάστη, η Ευρωδίκ και το Συνορέξ. Πρέπει να έχουν αυξηθεί οι δικαιοδοσίες τους τα τελευταία χρόνια και μερικές φορές ξεπέρασαν και την αρχική τους εντολή. Επίσης, τους έχουν δοθεί ορισμένα σοβαρά καθήκοντα, δηλαδή δυνατότητα παρέμβασης ακόμη και στα κράτη-μέλη. Εγώ είμαι μεταξύ εκείνων των περισσότερων στο Κοινοβούλιο που υποστηρίζουν την αύξηση αυτών των δικαιοδοσιών των υπηρεσιών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Δηλαδή την εφαρμογή της ε, στρατηγικής εσωτερικής ασφαλείας της Ένωσης που ταυτίζει τους πέντε κύριους κινδύνους ε, οργανωμένο έγκλημα, κυβερνοέγκλημα, τρομοκρατία, διαχείριση κρίσεων και ασφάλεια γενικότερα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και περισσότερη εποπτεία. Η ενδυνάμωση της εντολής του Frontex συζητήθηκε το Σεπτέμβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναγνωρίστηκε εκεί η ανάγκη να υπάρχει πιο γρήγορη ανταπόκριση στα προβλήματα της μετανάστευσης ιδιαίτερα βάσει των τελευταίων εξελίξεων στη Μεσόγειο. Όπως ξέρετε από τις αρχές του χρόνου έχει γίνει τεράστια κίνηση πληθυσμών στις χώρες της Βόρειας Αφρικής πράγμα το οποίο ε, δοκίμασε ιδιαίτερα τα συστήματα υποδοχής που έχουμε και από, την, και από το Σέγγεν και γενικότερα στην Ένωση και χρειάστηκε η κινητοποίηση πολλών όλων των ευρωπαϊκών χωρών και η χρησιμοποίηση όλων των χρηματοδοτικών και διοικητικών εργαλείων που διαθέταμε. Η, δια... η ενίσχυση της Σενγενική διακυβέρνησης είναι κάτι ουσιώδες αν θέλουμε να παίξουμε σοβαρά το ρόλο μας ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και να οικοδομήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο νέος αξιολογικός μηχανισμός του Σένιγκεν θα είναι τμήμα μέρος της ανταπόκρισης που χρειάζεται για το πρόβλημα αυτό γιατί θα παρατηρεί, θα επιτηρεί οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης των συνόρων και θα διασφαλίζει αποτελεσματικό έλεγχό τους από κάθε χώρα μέλος. Η, το δε Frontex θα παίζει όλο και περισσότερο ρόλο όχι μόνο για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ή λαθρομετανάστευσης, αλλά επίσης θα βοηθάει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα για τις μεταμέτρες μεταναστευτικές ροές. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί όμως ότι αυτή η νέα εντολή του Frontex σημαίνει επίσης και ότι υπάρχουν και ορισμένοι κίνδυνοι, δηλαδή ο ιδιωτικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των προσωπικών δεδομένων είναι πρόβλημα. Πρέπει να, δεν έχουμε ακόμη βρει ποιο είναι το καλύτερο σύστημα που να διασφαλίζει και την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ακόμη και αν σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας ο πρώην τρίτος πυλώνας έχει καταργηθεί, παρόλα αυτά πρέπει να καταπολεμήσουμε την τάση να διατηρείται αυτός ο τρίτος πυλώνας από αδράνεια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το θέμα αυτό των μεταναστευτικών ροών και του ελέγχου στα σύνορα ε, είναι κάτι που αφορά κεντρικά το θέμα της εθνικής κυριαρχίας του κάθε κράτους που είναι ακόμη ο μόνος υπεύθυνος για τον έλεγχο στα εξωτερικά του σύνορα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας στο γεγονός ότι χρειάζεται και μια ευρωπαϊκή πολιτική για όλα αυτά, πράγμα που φάνηκε καθαρά τα τελευταία χρόνια και κάθε φορά όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα εθνικά αναγνώριζαν ότι υπάρχουν, έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές που είναι πια, καθιστούν πια τις κινήσεις αυτές και τους ελέγχους στα σύνορα το πιο ορατό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τελειώνω υπενθυμίζοντας ότι ο αριθμός των ευρωπαϊκών υπηρεσιών έχει αυξηθεί στις 10. Το Κοινοβούλιο μπορεί να αρκεστεί στον υπάρχοντα προϋπολογισμό ή πρέπει να προβλέψει νέους τρόπους χρηματοδότησης ίσως από το ετήσιο πρόγραμμα που θα καθορίζεται κάθε φορά για τις δραστηριότητες των υπηρεσιών. Έχουν γραφτεί διάφορες γνωμοδοτήσεις και ακουστεί ότι δεν χρειάζεται καμία αύξηση. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ. Είναι ουσιώδες να υπάρξει πραγματική δημοκρατικός έλεγχος των δραστηριοτήτων τους. Ιδιαίτερα θέματα δοσιλογίας ευθύνης, λογοδοσίας εννοώ, ευθύνης και ελέγχου προστασίας ημί των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το διαθεσμικό παιχνίδι δεν αρκεί. Πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες ε, διάδοσης των πληροφοριών, της δημιουργίας δικτύων, σύνδεσης των εθνικών κομμάτων με το ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεννόησης των εισηγητών που έχουν παρεμφερεί θέματα. Νομίζω ότι στα εθνικά σας κοινοβούλια πρέπει να ορίσετε υπεύθυνους ε, επιτήρησης των διαφόρων ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Ο πρόεδρος Λόμπ Αγγιλάρ πριν από λίγα λεπτά μίλησε και αυτός για την ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων για την αξιολόγηση των εργασιών των υπηρεσιών αυτών. Τέλος, κυρίες και κύριοι φουλευτέ, χρειάστηκαν 50 χρόνια για να πραγματοποιηθεί η εσωτερική αγορά. Αλλά μόνο 12 χρόνια ασχολούμαστε για τη δημιουργία του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης κτλ. Κινούμαστε μεν προς τη σωστή κατεύθυνση μέσω της συγγραφής της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της συμπερίληψής της στη συνθήκη, αλλά στη μεταβατική αυτή φάση που ζούμε θα ήταν λάθος ή και επικίνδυνο να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη ασφαλείας χωρίς διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία. Από εμά όλους εξαρτάται με την επικοδομητική μας συνεργασία να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις που εκφράσατε. Και να πω ότι όταν η δική μου επιτροπή στον Οικοτολόνο κατάρτιζε την εκθεσή τη για τι στρατηγικέ εσωτερική ασφάλεια, είχαμε ένα πολύ καλό διάλογο με την κυρία Μπορσελίνο, που είναι η συγγήτρια στην Επιτροπή Λίμπη για το θέμα αυτό. <laughs> Και νομίζω ότι αναγνωρίζουμε πως αυτό ήταν ένας από τους τρόπους με τα οποία τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεργαστούν. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σα, λοιπόν ο κύριο Κίδας από το Κοινοβούλιο της ε, Μεγάλης Βρετανίας θα είναι επόμενος Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε την Προεδρία εδώ, Λόρδε Χάνη, Ένα από τα πολύ θετικά των οργανωμένων συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση απόψεων ε, και εγώ μπορώ να συμφωνήσω και να διαφωνήσω με διάφορους. Ε, τώρα εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε ο Κάρλος, ο συνάδελφος από την Πορτογαλία. Έχει απόλυτο δίκιο σε όσα λέει για την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερο έλεγχο Γι' αυτό είναι το σημείο αφετηρίας μου. Μου υπενθύμησε ότι ε, ξεκίνησε ε, στο Τάμπερε και εγώ μπορώ να σου πω ότι εγώ εκεί παρευρύθησα την πρώτη φορά ε, σε ε, συνεδρίαση ως υπουργό αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Με είχε διορίσει ο κύριος Μπλερ και πρώτη φορά παρευρέθησα σε τέτοια συνεδρίαση όμως ε, μπορώ να σας πω ότι διαφέρουν οι καιροί από τότε σε σχέση με το πώς εξελίχθηκε η στρατηγική τα τελευταία 10-11 χρόνια και ε, από ό,τι φαίνεται έχουμε τώρα ένα ρόλο που περισσότερο εφαρμογή παρά συντονισμού και πρέπει να είμαι προσεκτικό για τον συνάδελφο Κλίβιν Χόπκιν που προέρχεται από ε, την ε, Επιτροπή Ελέγχου του Κοινοβουλίου. Έχει διαφορετικέ απόψει από μένα, αλλά κάτι που μα ενώνει όλου στην αίθουσα είναι η ανάγκη για τον κατάλληλο και τον ορθό έλεγχο. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστά όσα υπόθηκαν από τον Κάρλος και Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε πρακτικά θέματα. Τι κάνει η δική μου επιτροπή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για να προσπαθήσει ε, να κάνει αυτούς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να λογοδοτήσουν. Έχουμε διάφορες ε, μεθόδους εργασίας. Ο τρόπος που εργάζεται η Επιτροπή Συντορικών Υποθέσεων στο Βρετανικό Κοινοβούλιο είναι να βασίζει όλα όσα κάνουμε σε αποδείξεις που καταφτάνουν ενωπιών μας. Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα κάνουν και οι συνάδελφοι σε άλλα κοινοβούλια. Αλλά επίσης σκέφτομαι ότι ένα ουσιαστικό τμήμα των όσων μπορούμε να πετύχουμε ως προς ε, τη διαφάνεια και τον έλεγχο είναι να έχουμε άμεσες επαφές ε, με συναδέλφους σε άλλα κοινοβούλια στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Γι' αυτό χθε συναντήθηκα με τον ε, Προεδρό της Επιτροπής Ιστορικών Υποθέσεων του Γαλλικού Κοινοβουλίου. Την επόμενη εβδομάδα έχω άλλη μια συνάντηση με συναδέλφους ε, σε, από άλλο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν λίγε εβδομάδε, ολόκληρη η Επιτροπή Ιστορικών Επιθέσεων μετέβη στην Ελλάδα όπου ε, συναντήσαμε τους ε, εταίρου μα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μάθαμε κι εμεί και ακούσαμε τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά σύνορα και πρέπει φυσικά ως ε, ένα βαθμό να ερχόμαστε εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αυτό είναι το κύριο όργανο που ελέγχει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς δεν, ε, εμείς ε, όλοι προερχόμαστε, ε, που προερχόμαστε από τέτοιες επιτροπές που έχουν ένα ρόλο ελέγχου, δεν θα πρέπει να περιμένουμε, δεν θα πρέπει να έρθουν αυτοί οι οργανισμοί να, από μόνοι τους να καταθέσουν αποδείξεις ενώπιόν μας Παραδείγματο χάρη, είχαμε το διευθυντή τη Europol να έρθει στο Λονδίνο για να απαντήσει ε, για τη δραστηριότητα τη Europol. Όπω ε, ξέρετε, όλοι αντιμετωπίζουμε οικονομικέ δυσκολίε και δεν μπορούσαμε να πάμε στη Βαρσοβία. Είναι πολύ περιορισμένε οι δυνατότητε επισκέψεων των βουλευτών. Έτσι λοιπόν πρέπει να διαλέγουμε πάρα πολύ προσεκτικά που πηγαίνουμε. Όμω ε, μπορέσαμε με τηλεδιάσκεψη να συζητήσουμε με τον ε, διευθυντή της Frontex ε, και μπορέσαμε να έχουμε άμεση επαφή με τη Frontex, όπως σας είπαμε βιντεοδιάσκεψη, ε, και να ρωτήσουμε τι συνέβη στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έχει δίκιο ο Κάρλος. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά όργανα, όμως ένα από τα προβλήματα που έχουμε εμείς ως βουλευτές είναι ότι έχουμε ε, την δυνατότητα να ελέγξουμε ορθά αυτούς τους οργανισμούς. Φυσικά έχουμε συζητήσει τη Europol, τη Frontex, ε, ξέρουμε ότι και Είσαι και κάνει δουλειά σε ό,τι αφορά ε, τη στρατηγική ασφαλεία και θέλω να μεταβώ στη Λιόν για να συναντήσω του συναδέλφου στην Ιντερπολ. Γιατί ένα τμήμα τη δουλειά που κάνουμε έχει να κάνει με την εμπορία ανθρώπων και δεν ε, σταματά απλώ τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η προηγούμενη συζήτηση που είχαμε εδώ για, για τη Frontex. Δηλαδή, ε, όταν ε, περάσουν ε, κάποια τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ αργά. Ακούσαμε τι είπε και η Ελληνίδα συνάδελφος, ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι χώρες προέλευσης των λαθρομεταναστών και ε, πηγέ εμπορία ανθρώπων. Έτσι λοιπόν πρέπει να τα δούμε και αυτά τα θέματα αν θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματο και τη λαθρομετανάστευση ε, και τη εμπορία ανθρώπων. Όταν επισκεφτήκαμε στην Ελλάδα, μιλήσαμε με τους ανθρώπους που ήταν υποκράτηση και ακούσαμε ότι πολλοί από αυτούς είχαν έρθει από το Αφγανιστάν, από το Ιράν, είχαν ε, ταξιδέψει, είχαν ε, περάσει όλη την Τουρκία ε, και μάλιστα πολλοί από αυτούς είχαν πληρώσει 5.000 ευρώ ο καθένας για να μπουν στην Ελλάδα. Και πιθανότατα μετά θα φτάσουν στο Λονδίνο, στο Άμυντο, στο Παρίσι και σε άλλες χώρες ακόμη και στη Λισαβόνα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτόν τον έλεγχο και είναι σημαντικό εμείς ε, να ακούμε τους εκπροσώπους αυτών των οργανισμών. Πολύ συχνά ε, υπάρχει ένα θέμα που κυρίως ε, αφορά ε, δύο κοινοβούλια ή περισσότερες, εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε να συναντούμε τους συναδέλφους για να είμαστε σίγουροι ότι κάποιοι διευθυντές ε, παρουσιάζονται να λογοδοτήσουν σε κάποιες κοινέ συνεδριάσεις. Ε, χτες ε, πρότεινα ε, στο συνάδελφό μου, στον ομολογό μου από το Παρίσι, να μεταβούμε στο Αφγανιστάν και να εξηγήσουμε στον Βρετανό φορολογούμενο τι ακριβώς κάνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιστορικών Υποθέσεων στο Αφγανιστάν. Αλλά αν δούμε τη λαθρομετανάστευση, πολλά από αυτά ξεκινούν στο Αφγανιστάν. Τα εγκληματικά δίκτυα των ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων ξεκινούν από την Καμπούλ γιατί ε, εκεί ακριβώς ε, πληρώνουν οι άνθρωποι για να ε, περάσουν όλα τα σύνορα μέχρι να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση λοιπόν είναι πολύ σημαντική και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξή. Το που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους διαδικασίες είναι να προσπαθούμε, όταν μάλλον ε, επιζητούμε να λογοδοτούν αυτοί οι οργανισμοί, ε, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει follow-up, ότι υπάρχει συνέχιση. Πρέπει να ε, δίνουμε και κάποια ε, κριτήρια σύγκριση για αυτού του οργανισμού. Ε, Παραδείγματο χάρη, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε και την υπηρεσία συνόρων που είναι αρμόδια για ε, τη μετανάστευση. Ετήσια ο διευθυντή αυτή τη υπηρεσία παρουσιαζόταν σε εμά. Εκπονούσαμε έκθεση και τα τρία χρόνια μετά βλέπαμε την έκθεση και λέγαμε πείτε μα τι κάνετε τα τρία τελευταία χρόνια. Τώρα αλλάξαμε προσέγγιση. Τώρα του θέτουμε συγκεκριμένε ερωτήσει στι 10 πολλέ τι αποκαλώ εγώ, αλλά έχουμε 50 μονομένε ερωτήσει που του ρωτάμε. Και στο τέλος κάθε τους ε, ε, βλέπουμε ε, αποφασίζουμε βάσει των τάδε 50 ερωτήσεων ότι θα ελέγξουμε ε, τον τάδε οργανισμό. Το κάνει το ίδιο το κοινοβούλιο, δεν το χρειάζεται να το κάνει η κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, ε, βάσει των συζητήσεων που έχουμε και με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να εκπονήσουμε 10-15 ερωτήσει κλειδιά και θα τι θέτουμε στη Europol και στου υπόλοιπου οργανισμού και να ξέρουμε ότι έχουμε κάποιο κριτήριο σύγκριση για το μέλλον. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ο τελευταίος ομιλητής, προτού προχωρήσουμε σε μια πιο γενική συζήτηση, η κυρία Λάμπερτ που είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μέλος της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε πρώτον γιατί καθυστέρησα αλλά είχαμε ψηφοφορίες όπου έπρεπε να παρίσταμε και δεύτερον διότι είμαι η τρίτη Αγγλίδα σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές ε, υπάρχει πολιτική ποικιλομορφία μεταξύ μας. Ε, είμαι υπεύθυνη εις ε, την Επιτροπή για την λειτουργία αυτών των οργανισμών και ε, ανέρχεται η αρχή αυτή σε μερικά χρόνια όταν προσπαθήσαμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσουμε τις επιδόσεις όλων των οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση ε, διότι βλέπετε ότι προσπαθώ να πω ότι όλα εξαρτώνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι όμως έτσι ε, βεβαίως αξιολογούμε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, εις ε, την, ε, τον αναλυτικό φάκελο 32 στο πακέτο που σας δόθηκε αναφέρονται εδώ ο, εξετάζουμε τις αρμοδιότητες των διευθυντών τον τρόπο λογοδοσίας τις, τις δημοσιονομικές πτυχές και την δημοκρατική λογοδοσία Γι' αυτό και πιστεύω ότι τα πορίσματα αυτών των συνεδριάσεων θα είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να αξιολογηθούν από την ε, αρμόδια ομάδα εργασίας. Διότι αισθανόμαστε πολλές φορές, όπως είπε και ο κύριος Κοέλιο, ότι ζούμε ε, σε κάποιο παρελθόν και τώρα είμαστε εντός ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν πρέπει απλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι το πηλίκον των μερών αλλά να υπάρχει και μία λεπή δραστηρία κοινοβουλευτική σχετικά με ε, την εποπτεία διότι στο παρελθόν ένα πρόβλημα υπήρχε με τη λογοδοσία διότι βλέπαμε ότι ε, όταν λειτουργούσαν οι διάφοροι οργανισμοί υπήρχαν κάτι ασαφείς περιοχές που δεν ανήκαν σε κανέναν και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σε μια δημοκρατία διότι αρχίζει να υπάρχει μια επέκταση ορισμένων οργανισμών τους οποίους κανείς δεν παρακολουθεί και κανείς δεν εποπτεύει. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι οργανισμοί τώρα έχουν όλο και περισσότερους ρόλους που αναλαμβάνουν σε σχέση με τις τρίτες χώρες, ιδίως ε, τις, τους οργανισμούς στηρίξεως ε, του ασύλου. Έπρεπε να δούμε ε, γι' αυτό πού θα τοποθετηθούν τα όρια και ε, ποια θα ήταν η νομοθεσία η οποία θα έπρεπε να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί. Ε, ποιες είναι οι πράξεις ε, οι οποίες έπρεπε να νομοθετηθούν και να εφαρμοστούν. Όλες αυτές οι πράξεις όμως έχουν μία πολιτική διάσταση και για την Frontex είδαμε ε, ότι υπάρχει μία διάσταση ασφαλείας σχετικά με τα σύνορα, θέματα τα οποία γνωρίζετε, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και διασυνδέσεις με άλλους οργανισμούς, εκ των οποίων η μία έχει σχέση με τη Frontex, δηλαδή κατά πόσον επικαλύπτεται με το ΝΑΤΟ. Πώς λοιπόν διακρίνεται ε, την ε, ε, λογοδοσία σε αυτό το τομέα διότι αν υπάρχει ασάφεια στη λογοδοσία υπάρχει ασάφεια και στην ανάληψη ευθυνών. Δηλαδή κανείς δεν έστειλε κάποια ελικόπτερα κάπου. Εάν δηλαδή προσπαθείτε εσείς να εντοπίσετε τι προκάλεσε κάποια ενέργεια και ποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξαμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε, κοιτάξαμε όλα αυτά τα πρακτικά προβλήματα και ε, δεν ξέρω εάν ο πρόεδρος που τώρα παρακολουθεί κάποιες πληροφορίες ε, κοίταξε, τι, σας είπε τι κάναμε στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υποθέσεων. Ε, τα απορίσματα παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα ή στην Επιτροπή Ελευθεριών και εξετάσαμε τους διάφορους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να δούμε πόσο ε, πρέπει να συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και ε, ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια γίνονται χωριστές μελέτες και θα διατυπωθούν χωριστά ψηφίσματα αλλά τονίσαμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και τα μέτρα αυτά να προλαμβάνουν τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν σε ορισμένους οργανισμούς. Υπήρξε μία μελέτη σχετικά με την εποπτεία των οργανισμών πληροφοριών που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Ελευθεριών και το Κοινοβούλιο αλλά δεν είμαστε υπέρ μίας δια κοινοβουλευτικής επιτροπής όπως αυτή την οποία προωθούσε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, έχουμε προτείνει ένα μόνιμο διακοινοβουλευτικό οργανισμό σε μόνιμη επαφή με αυτούς τους οργανισμούς και με επιτροπής όχι μόνο του ε, ε, ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και άλλες και ε, να υπάρχουν και οι αρμόδιοι εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων κοινοβουλίων που θα συμμετέχουν, να υπάρχουν εμπιστευτικές ομάδες εργασίες οι οποίες θα συζητούν τα διαβαθμισμένα προγράμματα, τη συνεργασία με τρίτες χώρες και άλλα θέματα κατά τρόπον ώστε να δούμε την αναλογικότητα του τι συμβαίνει από πλευράς δημοσιονομικής διότι χωρίς προϋπολογισμό σε κάθε δεύτερη γραμμή δεν μπορούμε να διατυπώσουμε τίποτα. Και ένα άλλο θέμα που απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι οργανισμοί αυτοί τουλάχιστον ε, συμβολικά ορισμένες ενέργειες για να αποδείξουμε ότι κάτι συμβαίνει και αν θεωρείται ότι είναι αναλογικό και αποτελεσματικό. Αυτό το οποίο ακούμε λοιπόν για, το κοινοβούλ, για τις ανταλλαγές μεταξύ κοινοβουλίων ε, είναι πολύ σημαντικό και η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι τακτική αλλά και οργανωμένη μεταξύ των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θα υπάρχουν δηλαδή τα ε, περίφημα σημεία επαφής όπως τα λέμε στην Ευρώπη ή αν υπάρχει κάποιος τρόπος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε τάσεις οι οποίες μας ανησυχούν γιατί κάτι που ανησυχεί τη Δανία ανησυχεί και την Πορτογαλία θα έπρεπε ίσως να το εξετάσουμε ε, πιο διεξοδικά και το ίδιο συμβαίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά θα μας βοηθούσαν. Θα μπορούσαμε να να βοηθηθούμε από την επιχειρησιακή εποπτεία που εξασκούν τα εθνικά κοινοβούλια και ε, ε, η Επιτροπή Ελευθεριών είναι υπεύθυνη για να προβαίνει σε πιο συστηματοποιημένη εποπτεία και ε, υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν επαφές με τα Εθνικά Κοινοβούλια διότι δεν είναι μόνο θέμα ε, εσωτερικών υποθέσεων όταν μιλάμε για ασφάλεια και για λαθρομετανάστευση υπάρχουν θέματα στα οποία άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων και γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε την εργασία των διαθεσμικών ομάδων εργασίας να σκεφτούμε και να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει μία παρακολούθηση και ενημέρωση μετά τις συνεδριάσεις και όχι απλώς μία τυχαία συγκέντρωση ερωτήσεων και θεμάτων γιατί ο καθένας πρέπει να κάνει μία ερώτηση διότι διαφορετικά δεν αισθάνεται ότι έχει συμμετάσχει. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον όλα αυτά να οργανωθούν κάπως καλύτερα για να μπορέσουμε να επιλύσουμε βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις και έχουν σημασία για την οργάνωση των πολιτών και πέραν των εξωτερικών συνόρων. Ευχαριστώ. Και τώρα Φτάνουμε στο τέλος των ομιλητών και θα γίνει μια συζήτηση σύμφωνα με τους υιοθετημένους κανόνες, δηλαδή δύο ομιλητές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ένας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δύο λεπτά. Ε, εάν κάποιος θέλει να μιλήσει πέραν των εγγεγραμμένων, πέστε μου ούτε το. Καταρχώς, καταρχήν δίνει το λόγο στον εκπρόσωπο του Φινλανδικού Κοινοβουλίου. Ε, Κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο γιατί νομίζω ότι είχαμε δύο αποτελεσματικές ε, ημέρες συζητήσεων και ε, σαν μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτική εποπτεία των πράξεων που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόληψη του εγκλήματος και θα πρέπει να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ των μέτρων που προστατεύουν τους πολίτες αλλά και την, την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Παρακολουθούμε την την Europol και την Eurojust ε, και βλέπουμε ότι στη διαδικασία αυτή θα πρέπει ε, να ε, συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια και θεωρούμε ότι μία κοινή διαδικασία θα πρέπει να καταρτιστεί για την κοινοβουλευτική εποπτεία της Europol και Eurojust με ένα κοινό χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να υπάρχει απλή, σύντομη και συγκεκριμένη εποπτεία, δεν χρειαζόμαστε νέους οργανισμούς που να παρακολουθούν αυτές τις διαδικασίες αλλά υπάρχει το πρόσφατα ιδρυμένο διακυβερνητικό φόρουμ και ε, όπου συμμετέχουν και τα 28 σώματα άρα πρόκειται για όντως ένα κοινό οργανισμό 27 εθνικά και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εγκαίρως ε, την τεκμηρίωση διότι το να λάβουμε χθε το μεσημέρι ένα βουναλάκι ε, χαρτιών δεν βοηθάει διότι δεν προλαβαίνεις καν να δεις ποιο είναι το περιεχόμενο Νομίζω όμως ότι ε, υπάρχει ένα βασικό έγγραφο που είναι η πολυετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την λειτουργία της Europol και θα πρέπει να παρακολουθούμε τις στρατηγικές. Το Σουηδικό Κοινοβούλιο λοιπόν ε, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό, ένας κοινός οργανισμός οργανισμός ο οποίος θα συζητά τις στρατηγικές της Europol και της Eurojust. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μάργαρετ Μπορ από τη Γερουσία της Ολλανδίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που παρευρίσκεστε εδώ και για τη συζήτηση αυτή. και νομίζω ότι η συζήτηση θα ήταν καλύτερη αν είχαμε προετοιμαστεί καλύτερα. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές δηλαδή και αν εστιαζόμασταν περισσότερο στα πραγματικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε γιατί ναι, μεν λαμβάνουμε πολλέ πληροφορίε και υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Υπήρξε μια ανταλλαγή δηλώσεων, αλλά στη συνέχεια τι θα γίνει. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούμε για την επόμενη φορά να εστιάσουμε κάπου περισσότερο για το θέμα της λογοδοσίας των οργανισμών. Υπήρξαν κάποιοι ομιλητές που επικεντρώθηκαν στο εθνικό τμήμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτά, δηλαδή να καλούμε τους διευθυντές των οργανισμών στην εθνικά κοινοβούλια, να υποβάλλονται εκθέσεις και επίσης για το πώς θα αυξηθεί η λογοδοσία μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα του κοινού ελέγχου ουσιαστικά είναι κάπως απογοητευτικό το ότι δεν κάναμε ένα βήμα παραπέρα και δεν είχαμε μια πραγματική συζήτηση από αυτού. Γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικό και θα πρέπει να συζητηθεί περισσότερο εις βάθος. Δηλαδή πώς θα έχουμε ένα ενδιαφέρον βήμα που θα λειτουργεί. Και ελπίζω ότι η συνέχιση αυτής της συζήτηση δεν θα είναι ότι την επόμενη χρονιά θα κάνουμε την ίδια διάσκεψη, αλλά θα σημειωθεί πρόοδο. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο ε, το λόγο πριν να δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ για να απαντήσουν. Έχουμε λίγο χρόνο αν επιθυμείτε το λόγο. Αλλιώς θα προχωρήσουμε στα μέλη του πάνελ. Δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Um, Μάλιστα. Στα αντίστροφα από τα αριστερά μου, συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι και δύο μιλητές από Σουηδία και κατοχώρες ανέφεραν την ανάγκη για συνέχιση δηλαδή η ανταλλαγή των πληροφοριών πριν από τέτοιε εκδηλώσει. Πολύ ωραία να ερχόμαστε στι Βρυξέλλε, αλλά καλό είναι να έχουμε και λεπτομερεί πληροφορίε εκ των προτέρων. Και δεύτερον, η ανάγκη για συνέχιση μετά τη συνεδρίαση αυτή. Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμ, κάποιες εργασίες ε, ε, στις επιτροπές μας και θα ζητήσω από την πληθυσμό να πάνε ε, στις ιστοσελίδες των κρατών μελών που συμμετείχαν για να μάθει ε, τι ακριβώς έρευνες διεξάγεται. Εγώ μπορώ να σας πω στις δική μας, επιτροπή, δική μας επιτροπή κάνει μια έρευνα για τον εξτρεμισμό, δηλαδή γιατί κάποιοι πολίτες γίνονται εξτρεμιστές και επίσης κάνουμε και μια έρευνα για το hacking των τηλεφώνων. Θα το έχετε ακούσει. Αλλά δεν ξέρω αν ε, ο κύριος Χόπκινς ε, που ήρθε μαζί μου ε, από τον Ηνωμένο Βασίλειο θα ξέρω και το Επιτροπή τι ακριβώς ερευνά και είναι στην αίθουσα δίπλα μου, στη διπλανή πόρτα. Έτσι λοιπόν, αν και μου αρέσει η ιδέα ότι κάποιος από την Επιτροπή της κάποιος ίσως ο αντιπρόεδρος να μπορεί να λειτουργεί ως σημείο επαφής, είναι εξαιρετική ιδέα αυτή. Νομίζω ότι τίποτα δεν μα εμποδίζει παρόλα αυτά αύριο να πάμε στα εθνικά μα συνοβουλία και να ζητήσουμε από τι βοηθείε μα να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα του ζητήσω από τον βαθό μου να δει ε, τι ερευνάτε εσεί στι χώρε σα. Γιατί αν δούμε ότι κάνετε και εσεί κάτι που κάνουμε και εμεί γιατί η Europol, παραδείγματο χάρη, όπω είπαν και κάποιοι συνάδελφοι, καλό είναι να ανταλλάξουμε αυτέ τι πληροφορίε, να μην έχουμε επικαλύψει και αν έρθει ο διευθυντή τη Europol ή ο διευθυντή τη Frontex ενωπιών μα, ευχαριστώ να στείλω ένα email, δεν είμαι στο facebook και ούτε στο twitter, είμαι πολύ μεγάλος ε, για τα πράγματα αυτά, θα είναι ένα καλό παλιωμοβίτικο email. <laughs> Μας είπατε ότι ούτε εσεί, Στην Ουγγαρία μάλιστα μπορούμε τέλο πάντων να έρθουμε σε εύκολη επικοινωνία μεταξύ μα και να ενημερώσουμε ένα τον άλλο για το τι κάνουμε αν υπάρχει μια κοινή απειλή. Εγώ δεν ε, θα ήθελα να φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται σε επαφή μόνο με τις Ηνωμένε Πολιτείες για ιστορικούς λόγους ε, και υπάρχει και αυτή η προκατάληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ε, μετέβη στην Ουάσιγκτον και έμαθα ότι ένας συνάδελφος στην Ουάσιγκτον εκεί έκανε ακριβώς την ίδια έρευνα που κάνουμε κι εμείς για τον εξτρεμισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση. Και μου έδωσε τελικά ο συνάδελφο τι πληροφορίε αυτέ. Έτσι λοιπόν ευχαρίστω να το κάνουμε και με του Ευρωπαίου εταίρου μα. Και εν τω μεταξύ η Engine θα μπορούσε να δώσει μια συνέχιση σε αυτό το θέμα του διορισμού κάποιου αντιπροέδρου με επαφή. Πολύ καλή εξέλιξη. Είχαμε και μία διάσκεψη στο Λονδίνο για την εμπορία ανθρώπων. Πολλοί συνάδελφοι ήρθαν από τι ε, διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα άλλο τρόπο να λειτουργήσουμε. Αν κάποια ε, επιτροπή δική μα ε, ασχολείται με κάτι συγκεκριμένο, μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτήν εδώ και να σα πω ότι δεν επικεντρωνόμαστε στη Europol, αλλά αν κάποιο από εσά ενδιαφέρεται για τη Europol, ευχαρίστω να στείλω ένα μέλο τη δική μου επιτροπή στη χώρα σα, προκειμένου να συμμετάσχει σε μία τέτοια διάσκεψη. Νομίζω όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε, τόσο καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κοέλιο. Σας κατευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ συμμερίζομαι αυτά που είπατε ως προς το τι πρέπει να δώσουμε ως συνέχεια. Μάλιστα εχθές είπα σε μερικούς συναδέλφους σε ιδιωτικές συζητήσεις αυτό το πράγμα φτάνουμε στο τέλος της συνάντησής μας με την ιδέα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα καινούριο. Αυτό είναι τρομερό. Αλλά αυτό που επί το οποίο συμφωνούμε είναι ότι θέλουμε να συνεργαστούμε τα εθνικά κοινοβούλια με το ευρωπαϊκό. Οι συντονιστές μας συμφώνησαν να έχουν μία ειδική συνεδρίαση του Προεδρείου της Επιτροπής μας για να κάνουμε την αξιολόγηση αυτής της συνάντησης και να αποφασίσουμε τη συνέχεια. Και ο Πρόεδρος Αγγελάρ έκανε μία πρόταση σχετικά, δηλαδή να υπάρξει μία κοινή διαδικασία αξιολόγησης της δουλειάς των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Νομίζω ότι σε λίγο θα το ακούσετε και πιο επίσημα, γιατί όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας είναι καλό και οι εθνικοί βουλευτές να συμμετέχουν σε αυτές τις αξιολογήσεις αλλά πρέπει να υπάρξει μια κοινή διαδικασία αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα και ελπίζω η πρόταση του Προέδρου Λόπης Ζαγκυλάρ να εφαρμοστεί και έτσι θα υπάρξει αυτή η κοινή διαδικασία αξιολόγησης της δουλειάς των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας εκτιμά και αυτό στα συμπεράσματα, μερικά από τα συμπεράσματά μου είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε καλύτερα τους συναδέλφους για να ξέρουμε σε ποιον μιλάμε κάθε φορά. Η διαδικασία αυτή προσκλήσεων και λοιπά και οι τακτικών συναντήσεων είναι τελείως ουσιώδης. Για να μην υπάρχουν χωριστές συναντήσεις των εθνικών με τους ευρωπαϊκούς βουλευτές. λείπει αυτή τη στιγμή κάποιος διάλογος μεταξύ μας ενώ έχουμε κοινή ευθύνη αξιολόγησης. Τι να γίνει για την επόμενη φορά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε μερικά από τα κέρια ερωτήματα που να τα θέσουμε εκ των προτέρων πριν γίνει η συζήτηση για να ετοιμαστεί και η τεκμηρίωση θα ήταν πολύ χρήσιμο. Τουλάχιστον να διαβάσουμε ορισμένες συνόψεις πριν δούμε τα πλήρη έγγραφα. Πρώτα όμως να καθορίσουμε ποια είναι τα κέρια ερωτήματα, τι προτεραιότητες έχουμε, τι θα ενδιέφερε όλους. Ίσως να δημιουργήσουμε και καμιά ομαδούλα εργασίας για να τα καθορίσει αυτά. Έτσι θα ήταν καλύτερη η συνεννόηση μεταξύ μας για θέματα ασφαλείας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Φυσικά είναι βέβαιο ότι και άλλοι συμφωνούν με αυτές τις προτάσεις εδώ και νομίζω ότι έτσι οι συναντήσεις μας θα είναι πιο αποτελεσματικές. Να ξέρουμε φεύγοντας ότι «Α, ναι, αυτός ήταν ο σκοπός μας, αυτή είναι και η πρόταση». Είναι πιο ενδιαφέρον αυτό ως αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, υπήρχαν και άλλοι δύο μιλητές, αλλά ο ένας χρειάστηκε να φύγει γιατί έχει αεροπλάνο, ο δε πρόεδρος Αγγιλάρ έχει δουλειά με την Πολωνική Προεδρία. Και δεν θα είναι εδώ για το κλείσιμο. Πριν προσπαθήσω να συνοψίσω, έχω ένα τελευταίο αίτημα για παρέμβαση. Και αφού έχουμε χρόνο μπορώ να το δώσω στον κύριο Πάντζιο εκπρόσωπο της Τσεχίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τα οργανωτικά. Για την επόμενη συνάντηση θα ήθελα να έχουμε τα έγγραφα εκ των προτέρων. Αυτό είπε και η κυρία από τη Σουηδία. Γιατί έλαβα ένα τεράστιο όγκο γράφουν την τελευταία στιγμή στο γραφείο μου. Δεύτερον, είχα ένα ερώτημα, μια απορία στη συζήτηση για τα εσωτερικά σύνορα και δεν έλαβα απάντηση για να το πω ειλικρινά. Την επόμενη φορά ίσως να έχουμε δύο γύρους ερωτήσεων έναν πρώτο γύρο μετά να απαντούν οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών και μετά δεύτερο γύρο από τους, για τους εθνικούς βουλευτές ειδικά. Ίσως έτσι να είναι καλύτερη η συνεννόηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους και όλες και τους ομιλητές για τη συμβολή τους θα προσπαθήσω να βγάλω ένα-δυο συμπεράσματα. Αν και αναγνωρίζω ότι ως προσωρινός προεδρεύων σε μια οργάνωση 27 χωρών είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ικανοποιήσω τους πάντες. Πάντως αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσω νομίζω. Σημείωσα ότι στην τελευταία μας συζήτηση Υπήρξε μεγάλη σύγκληση απόψεων. Δεν άκουσα κανέναν να λέει ότι χρειάζεται κάποιο νέο όργανο ειδικά για αυτή τη δουλειά. Και η Βουλή των Λόρδων συμφωνεί απόλυτα, δεν χρειάζεται περισσότερη γραφειοκρατία. Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί και η εμπειρογνώμονες των οποίων τη γνώμη ζητήσαμε το ίδιο είπαν όχι απαραίτητο από την Επιτροπή Ελευθεριών αλλά όλοι όσοι μίλησαν. Απ' την άλλη άκουσα πολλούς να αντιδρούν σε αυτά που είπε ο πρόεδρος Αγγιλάρδη δηλαδή ότι η συνεδρίαση της επόμενης χρονιάς πρέπει να είναι πιο οργανωμένη, πιο αποτελεσματική, πιο ρεαλιστική από ό,τι πετύχαμε μέχρι τώρα. Αν και νομίζω ότι τις τελευταίες δύο μέρες κάναμε κάποια πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση, περισσότερη από τις προηγούμενες συναντήσεις, στις προηγούμενες συναντήσεις. Αυτό είναι ελπιδοφόρο, ελπίζω να μην έχει κανείς αντίρρηση. Ο πρόεδρος Αγγιλάρ πρότεινε να γίνει η επόμενη συνάντησή μας τον Οκτώβριο του 12 και ελπίζω ότι περισσότερα εθνικά κοινοβούλια βασιζόμενα στην σημερινή μας εμπειρία θα εκπροσωπηθούν διότι μου φαίνεται σαφές και εδώ συμφωνούν όλοι ότι για το θέμα αυτό που συζητήσαμε σήμερα και χθε και το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να παίξουν άμεσο ρόλο. Δεν υπάρχει κανένα, κανένα, καμία από τις δύο κατηγορίες που να έχει προτεραιότητα έναντι της άλλης, αλλά οι συνθήκες προβλέπουν ρητά ότι η κύρια ευθύνη για την εσωτερική ασφάλεια είναι των χωρών μελών. Όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω των δικαιοδοσιών που έχει συναπόφαση και στον προϋπολογισμό έχει και αυτό έναν σαφέστατο ρόλο. Επομένως το μόνο λογικό θα ήταν να συνεχίσουμε τις συναντήσεις μας με τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι εδώ έχουμε κοινή προεδρία από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών και κάποιον από τα Εθνικά Κοινοβούλια τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν δύο ευκαιρίες να μιλήσουν και το Ευρωπαϊκό μία κάθε φορά και αυτό σωστό και δεν υπάρχει θέμα πρωτοκαθεδρίας γιατί δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Έχουμε και η μεν και η δε τις ευθύνες μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά και η κάθε κατηγορία την εφαρμόζει τις ευθύνες της όπως νομίζει σωστότερο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο συλλογικοί. Αυτό ακούστηκε σαφώς από τη συζήτηση. Χρειάζεται απολύτως να υπάρξει μια συλλογή δεδομένων πριν από την οργάνωση της κάθε συνάντησης. Εχθές άκουσα τον Επίτροπο να λέει, την Επίτροπο να λέει ότι είχε σκοπό του χρόνου η ετήσια έκθεση για την Ευρωπόλ να διατεθεί εγκαίρως για να μπορεί να συζητηθεί στην τέτοια μας συνεδρίαση. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και για τις εκθέσεις περί των άλλων υπηρεσιών, την Ευρωπόλ και την Ευρωτζάστ, ώστε να έχουμε τα στοιχεία και το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια εγκαίρως και πάνω απ' όλα να τα έχουν όλοι όσοι έρθουν στη συνάντηση αυτή του χρόνου. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτά που είπε ο κύριος Αγκυλάρ και η Επίστροπος Μάλστρομ θα, θα εισακουστούν και θα οδηγήσουν σε κάποια σωστότερη ανταπόκριση των εκκλήσεων που ακούστηκαν ότι δεν είναι άχρηστο να έχουμε τεράστιους σωρούς εγγράφων την τελευταία στιγμή. Άλλη ιδέα που εξέφρασε ο κύριος Αγγελάρη ήταν ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συνεννοούνται με το ευρωπαϊκό και να του υποβάλουν ό,τι ιδέες έχουν για την καλύτερη διοργάνωση της δουλειάς αυτών των υπηρεσιών πριν γίνει η ετήσια συνάντηση. Είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον για τη δική μου επιτροπή θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην έκκληση αυτή και νομίζω ότι και άλλα εθνικά κοινοβούλια αλλά και το ευρωπαϊκό πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιο θα είναι το θέμα της συζήτησης πριν προσέλθουν οι συνάδελφοι. Τρίτον, προφανώς γιατί το είπαν όλοι, χρειάζεται ανάγκη μεγαλύτερης συνεννόησης μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού ως προς το τι έρευνες κάνουν, τι μελέτες αναλαμβάνουν για να μπορούν να ωφεληθούν οι μένα από, τις των ΔΕ να γνωρίζουν τι γίνεται στις κάθε, στην κάθε χώρα μέλος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να μην ξεπέρασα τα όρια της εντολής μου. Δεν μπορώ βέβαια να επιβάλλω σε κανέναν τίποτα, αλλά θέλησα απλώς να σας επαναλάβω μερικές από τις προτάσεις που έκανε ο πρόεδρος Αγγιλάρ. Θα τα μεταφέρω στη Βουλή των Λόρδων, ελπίζω και άλλα κοινοβούλια να μεταφέρουν τις ιδέες αυτές και ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι του χρόνου η συνάντησή μας να είναι πιο αποτελεσματική, πιο συστηματικά οργανωμένη και καλύτερα πεπληροφορημένη από ό,τι η φετινή. Αν το καταφέρουμε αυτό, τότε νομίζω ότι θα αρχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτά που μας επιβάλλει το άρθρο 88 της συνθήκης, δηλαδή σωστή κοινοβουλευτική εποπτεία μέσα στην καινούργια αυτή θεσμική δομή. Αν είναι όλοι ικανοποιημένοι λοιπόν με αυτά τα συμπεράσματα, ο κύριος Αγγιλάρ μου ζήτησε να κλείσω εγώ τη συνάντηση, ζητά συγγνώμη γιατί χρειάστηκε να φύγει, αλλά πρέπει να εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια συνάντηση με την Πολωνική Προεδρία και γι' αυτό δεν μπορούσε να λείπει από εκείνη τη συνάντηση. Θα ήθελα λοιπόν την απουσία του να τον ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους στη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να διοργανωθεί αυτή η συνάντηση και για όλα όσα έκαναν για να την πραγματοποιήσουν και ελπίζω να μπορέσουν να προωθήσουν τα πράγματα σε συνδυασμό με τις γραμματείες των Εθνικών Βουλών που είναι ισότιμοι εταίροι, όχι υποδεέστεροι. Για να δούμε αν του χρόνου δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά που ζήτησε ο πρόεδρος Αγγιλάρ και που όλοι θεωρούμε ότι θα συνέβαλαν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και όπως είπα λοιπόν κλείνω τη συνάντησή μας τώρα ευχαριστώντας ξανά την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών για όλα όσα έκανε για να πετύχει η εκδήλωσή μας. Σας κατευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση.